Ε, υπάρχουν προβλήματα με τα πρακτικά. Κυρίως ε, αναφέρομαι σε εκείνους που τα έχουν διαβάσει, βεβαίως. Κλείνει λοιπόν και το θέμα αυτό. Ερχόμαστε στα ζητήματα των ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Ε, οι διαπραγματεύσει στην ΑΦΕΤ ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και στην Επιτροπή ανάπτυξη τη Δευτέρα το βράδυ. Το ΚΟΡΕΠΕΡ συμφώνησε με όλες τις διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμα είναι έτσι και έτσι μου έγραψαν, μου διαβίβασαν μια μακροσκελή υποσημείωση για όλα αυτά και το συνοψίζω με το έτσι και έτσι. Λοιπόν, την, ε, η επιθυμία μας, το αίτημά μας μάλλον να περάσει μέσω κατεξουσιοδότηση πράξεων απέτυχε παταγωδόσα ε, και υπήρξε μία συνεργασία μεταξύ της γραφειοκρατίας των Βρυξελών και εθνικών ε, γραφειοκρατιών. Ε, κυρίως από την Κομισιόν ο συνάδελφος Φιούλε ε, βρίσκεται πίσω από αυτά και αυτό δίνει έναυσμα σε κάποιους προβληματισμούς. Βεβαίως είναι ένα πρόβλημα γενικής φύσεως σε σχέση με τον τρόπο εργασίας της Κορεπέρ. Υπάρχει ένας εντεταλμένος ο οποίος δεν γνωρίζει ακριβώς ε, ποια είναι η εντολή του ε, και ο οποίος θα πρέπει να προσαρμοστεί σε κάποιες ε, αποφάσεις γιατί ακριβώς η Κορεπέρ εργάζεται με ένα τρόπο που είναι εντελώς ασύμβατος με το κλασικό σύστημα του ενός δεύτερου σώματος. Και νομίζω ότι στη την νομοθετική διαδικασία αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αλλά θα πρέπει να πω ότι αν εξαιρέσουμε αυτό, πετύχαμε κάποια πράγματα όσον αφορά τα οριζόντια θέματα, καθώς και τις εκθέσεις που διαπραγματεύθηκαν οι συγητές, σημειώθηκαν κάποιες πρόοδοι. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους συγητές που πραγματικά έδειξαν μεγάλη υπομονή και ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι μπορέσαμε ε, μέσω παρακαμπτηρίων να πετύχουμε την προθεσμία των 3,5 ετών ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε ότι το βασικό μας επιχείρημα ότι δεν θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρως για 7 έτη, ε, το οποίο σημαίνει βεβαίως ότι το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να πει κάτι, να αναμειχθεί καθόλου σε αυτό το θέμα ε, στην επόμενη θητεία. Ε, όλα αυτά είναι κάπως ε, σύμβατα με την ε, δημοκρατικότητα ε, και ίσως η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής θα ήταν πολύ καλύτερη αν δεν υπήρχαν κοινοβούλια τα οποία διαταράσουν την πορεία, λένε ορισμένοι. Και αυτό πραγματικά είναι αστείο. Τώρα, όσον αφορά την επιστροφή των ροών ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον και νομίζω ότι μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε πολλούς ε, τομείς ε, που αφορά την κατανομή των κονδυλίων βάσει θεματολογικών ή γεωγραφικών δεξιών. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε μέσω των τροποποιηθήσεων κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Ε, πιο κάτω από το επίπεδο των κατεξουσιοδότηση πράξεων υπάρχουν τρόποι βάσει των οποίων μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα το Κοινοβούλιο. Τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τους συγητές να κάνουν συντομία κάποιες παρατηρήσεις ο κύριος Κούκραν για το εργαλείο της ε, γειτονίας. Παρακαλώ δύο λεπτά. Ε, μην μπείτε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες γιατί θα προκαλέσετε σύγχυση και θα παραπονδύσετε την ε, διενέργεια των εκλογών. Ευχαριστώ πολύ. Το κλειδί για τις διαπραγματεύσεις για το εργαλείο ε, γειτονίας ήταν πιο δημοκρατικό και κατά πολύ απλωστευμένο. Μετά από πολλές ε, συζητήσεις και διατύπωση κριτηρίων για τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού πετύχαμε συμφωνία για τα δύο βασικά τμήματα. Καταρχήν ε, μέχρι να τροποποιείται το φάσμα μέχρι 20% αλλά και να υπάρχει μια επιπρόσθετη υποστήριξη μόνο για εκείνες τις χώρες που έχουν ε, πετύχει προόδους στην, ε, στον εκδημοκρατισμό. Και αυτή η υποστήριξη θα εξασφαλιστεί ε, μέχρι το 10% του προϋπολογισμού. όσον αφορά ε, την ε, πρόοδο της βιώσιμης δημοκρατίας ως ε, μοναδικού κριτηρίου για τη χορήγηση υποστήριξης, κάτι το οποίο είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο, μπορέσαμε να εκπληρώσουμε αυτό το στόχο όλα αυτά εντάχθηκαν στο γενικότερο πλαίσιο χάραξης ε, πολιτικής. Στην αρχή το Συμβούλιο είχε κάποιες ε, αντιρρήσεις, αλλά τελικά μπορέσαμε να υποστηρίξουμε τις δικές μας ε, θέσεις. Όσον αφορά την ε, συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών, το τελικό κείμενο αντανακλά τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά το δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους του Κοινοβουλίου, διαπραγματευθήκαμε το παράρτημα όπως είχε τροποποιηθεί μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων που περιλαμβάνει τις βασικές προτεραιότητες και καταδεικνύει την, ε, ε, δίνει κάτι κατανομή των κονδυλίων. Ε, το 2018 θα υπάρξει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση ούτως ώστε το μελλοντικό κοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει αυτές τις ε, προτεραιότητες. Ε, αυτά τα είχαμε κατά νου στην αρχή της διαπραγμάτευσης με όρους των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά επιτεύχθηκε τελικά ήταν ακόμα πιο θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. López's tour is white. And up. Vielen Dank. Uh... Ah, no. Πώς θα δούμε ε, όσον αφορά το, όσον εργαλείο γειτονία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σκιώδη και όπως είπε ο Πρόεδρος θα ήθελα να τον συγχαρώ για την υπομονή που έδειξε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σε αυτό το δύσκολο έργο. Ε, οι οποίοι ήταν πραγματικά πιο υπομονετικοί από μένα τον ίδιο. Είναι σαφές ότι με αυτό το εργαλείο το οποίο προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας είναι μια νέα φάση ανάληψη εξωτερική δραστηριότητα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αρχή ενό νέου οικονομικού πλαισίου είναι αναγκαίο να συνοδευτεί αυτή η νέα φάση με ένα εργαλείο το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ε, πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω. Αυτό το εργαλείο είναι ο πρώτος, ο πρώτος του στόχος είναι η χρηματοδοτική υποστήριξη στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους στρατηγικούς μας εταίρους καθώς και η πολιτική ε, καθώς και η υποστήριξη πολιτικών, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις. Σε αυτό το κόσμο που όλα είναι όλο και πιο αλέντατα και όλο και πιο σύνθετα, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστική. Κατά συνέπεια, το εργαλείο αυτό θα μπορέσει να στηρίξει επίσης τη διεύρυνση της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Μπορέσαμε να τονίσουμε την ανάγκη το εργαλείο αυτό να συνεχίσει να υποστηρίζει προς τα έξω τις τρεις βασικούς στόχους αυτής της στρατηγικής που είναι όπως ε, γνωρίζετε και με αυτή τη στηρά αποσχόληση, καινοτομία, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και βιώσιμη ανάπτυξη. Στο μέτρο αυτό καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τις ε, επιχειρήσεις, ενεργειακή επάρκεια, βιώσιμη οικονομία, στήριξη προς την επιστήμη, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα κλπ. Επίσης θα προωθήσει την διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Επίση, την εξωτερική δράση είναι η προώθηση τη εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ολόκληρο τον κόσμο και ενίσχυση των δεσμών μα ε, με τους εμπορικούς μας εταίρους, σημαντικά στοιχεία αυτού του εργαλείου. Εξ ονόματος της Επιτροπής ΙΝΤΑ ε, διατυπώθηκαν κάποιες παράγραφες σε σχέση με το εξωτερικό εμπόριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντρικένεν που συνέταξε αυτές τις παραγράφους. Ε, το προσεχή Ιανουάριο θα ξεκινήσει το δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτή τη νέα φάση θέση ισχύ ε, του νέου εργαλείου ε, με ε, συναπόφαση του Κοινοβουλίου και άξιση πολιτικού ελέγχου έχουμε διατυπώσει τις ε, προτεραιότητες σε ένα παράρτημα το οποίο τροποποιείται βάσει των κατεξουσιοδότηση πράξεων ούτε ώστε ο νομοθετικός έλεγχος του Κοινοβουλίου καθώς και η αύξηση της συμμετοχής στη φάση του προγραμματισμού να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα αυτού του αργαλείου και ολοκληρώνω ζητώντας να υπερψηφίσετε αυτό το εργαλείο που θα βοηθήσει να προβάλλουμε και να ενισχύσουμε προς τα έξω τις αξίες και τα ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παρούσα συγκυρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσω για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το μέσο περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν πρόκειται μόνο γι' αυτό, αλλά πρόκειται και για το εργαλείο για την υποστήριξη της ε, δημοκρατίας. Πρόκειται για έναν από τους τομείς όπου η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη. Γι' αυτό λοιπόν από την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο πρέπει να το ερμηνεύσουμε συμπληρωματικά προς τα άλλα. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προαγωγή της δημοκρατίας ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλους τους τομείς και μόνο όπου δεν είναι δυνατόν να ε, παρακολουθεί κανείς ε, την πολιτική από άλλο πρίσμα, μόνο εκεί πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το εργαλείο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο και ο στόχος μας δεν ήταν να τροποποιήσουμε ουσιαστικά το μέσο αυτό, αλλά κατ' ουσία να εστιάσουμε την προσοχή μας σε εκείνες τις ε, προκλήσεις, ε, οι οποίες ε, αποδείχθηκαν νέε προκλήσεις. Αναφέρομαι στην Αραβική Άνοιξη και αναφέρομαι και σε άλλα σημαντικά θέματα, τα οποία μπορούν και αυτά να εξεταστούν κάτω από το πρίσμα του ε, μέσου μέσω αυτού περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο τρίτος ε, στόχος ε, τον οποίο εκφράζει αυτό το εργαλείο αλλά και αυτό εξετάζεται κάτω από το πλαίσιο της κοινή οδηγίας και του κανονισμού είναι οι θεσμικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά στον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για αυτό το εργαλείο, όλο και για όλα τα άλλα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει η περίφημη διάμεση αναθεώρηση και μάλιστα αυτή ε, να υπάρχει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το επόμενο κοινοβούλιο να μπορεί να επηρεάσει τα στρατηγικής φύσεως ε, θέματα κατά τη διαμόρφωση του εργαλείου. Δεν θα ήθελα τώρα να μπω σε λεπτομέρειες γιατί έχουμε μπροστά μας την ε, ψηφοφορία. Θέλω μόνο να σας πω ότι στις διαπραγματεύσεις τόσο με το Συμβούλιο όσο και με την Επιτροπή ε, πρέπει να στήσουμε για την ουσία, για την ισότητα των μειονοτήτων, για την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκονται, τη δύσκολη κατάσταση πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, για όλα αυτά επιτύχαμε συμφωνία και μάλιστα ε, χωρίς καθυστερήσεις. Λάμβαμε υπόψη μας και τα κοινωνικά δικαιώματα, το ανθρώπινο δικαίωμα για ε, σωστή και καλή διαβίωση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και το βασικό δικαίωμα να μπορεί κανείς να ε, ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, το Right to Conduct, a Business και αυτό έχει ενταχθεί στο εργαλείο για το οποίο συζητάμε. Όσον αφορά τις ε, κατεξοσιοδότηση πράξης, έχουμε ένα παράρτημα όπου περιλαμβάνονται οι πέντε βασικοί στόχοι του εργαλείου αυτό το ε, θέμα ε, θα ε, προσθετεί στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Στα οικονομικά δεν επιτύχαμε συμφωνία. Για πρώτη φορά λοιπόν αναφέρεται ότι οι παρακολουθήσεις εκλογών που χρηματοδοτούνται από το Μέσο περί Δικαιωμάτων δεν θα καταλαμβάνουν το 25% του προϋπολογισμού. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια συμφωνία η οποία άτυπα υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια και η οποία έλαβε πλέον μια καθαρά τυπική μορφή. Τελειώνοντας και νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον και κατ' ουσίαν επιβεβαιώνει και τη σημασία την οποία αποδίδουν όλοι σε αυτό το μέσο Μιλάμε για 1,3 δις ευρώ, για αύξηση κατά 20% στα μέσα που διατίθενται για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προαγωγής της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Λοχπίντα. Σήμερα ομιλώ εξ του εισηγητή μας, του κυρίου Πίτικοφερ, που δυστυχώς είναι άρρωστος. Επιτέλους έχουμε ένα τελικό εργαλείο, είναι το εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει στην σταθερότητα και την ειρήνη και θέλω να υπογραμμίσω κάποιες επιτυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Έχουμε την πρόληψη ε, συγκρούσεων ε, με οικονομική δραστηριότητα που διπλασιάζεται. Φτάνουμε σε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Από τις ε, πρόσφατες εμπειρίες μας σε χώρους όπως αυτούς που έλαβε χώρα η Αραβική Άνοιξη, η σταθερότητα ε, δυστυχώς ε, παραγώνισε την κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε ένα νέο τίτλο σε αυτό το μέσο που περιλαμβάνει και την ειρήνη και με τον τρόπο αυτό εκφράζεται καλύτερα ε, η προαγωγή της ειρήνης. Το εργαλείο το δικό μας έχει ως στόχο να βάλει τη συνεργασία όχι μόνο ανάμεσα κυβερνήσεις αλλά και ανάμεσα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι θα συνεχίσουν να ε, είναι το επίκεντρο των προσπαθειών μας. Η κοινωνία των πολιτών θα καθορίζει ρόλο ε, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Λόγω της ευαισθησίας που έχει η συνεργασία για θέματα που άπτονται της ε, ασφάλειας και αναφέρομαι κυρίως

σε μεταρρυθμίσεις έχουμε δημιουργήσει ένα μηχανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή αναγκάζονται να εφαρμόσουν ένα σύστημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό ως στόχο του ε, σχεδιασμού σε όλους τους τομείς. Επιπλέον, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να αναφέρονται στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του Μηχανισμού ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε ενισχύσει το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμπεριλαμβάνεται ο στρατηγικός διάλογος σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της εφαρμογής των δράσεων συμπεριλαμβανομένων και των κρίσεων. Έτσι λοιπόν ε, θα έχουμε μια πιο πλούσια μερίσια διάταξη, κυρίως στην ομάδα εργασία για την πρόληψη συγκρούσεων. Τέλος, θέλουμε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους και του κυρίου Πιτικόφερ, αλλά και εκ μέρους της κυρίας Μπρόντνα για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε με τους σκιοδησηγητές Γκαλτιέρη, Κίλα Λάμπστοφ και Λούζινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούτσεκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μιλάμε λοιπόν για την εκεί, βοήθεια και ε, είχαμε δυόμιση χρόνια σε βάθος διαπραγματεύσεων. Επιτεύχθηκε μια περιεκτική συμφωνία για το νομικό κείμενο για την ενίσχυση της ε, χρηματοδότησης. Μιλάμε ε, κατ' ουσίαν για μεγάλα ποσά που ξεπερνούν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά λοιπόν το Κοινοβούλιο συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία ως συνομοθέτης σε ίση βάση με το Συμβούλιο. Η, ε, ο συμβασμός που επιτεύχθηκε με τη Λιθουανική ε, Προεδρία είναι ρεαλιστικός και αντικατοπτρίζει βασικές προτεραιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε 4-5 προτεραιότητες. Δηλαδή, περιλαμβάνεται, ε, περιλαμβάνονται ε, γενικότεροι στόχοι ε, στο, πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης. Κατόπιν γίνεται λόγος για, τις, για τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας που ενισχύουν τον πολιτικό μας ρόλο στη διαδικασία της διεύρυνσης. Επίσης ε, ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό ε, να εφαρμοστούν οι στόχοι ε, και αυτό μέσα από τις αποκαλούμενες ε, θεματικές προτεραιότητες οι οποίες τροποποιήθηκαν από τις κατεξουσιοδότηση πράξεις μέσω πρόθεσμα. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο το νέο κοινοβούλιο θα έχει λέγει σε αλλαγές που μπορεί να προκύψουν τις προενταξιακές χώρες. Επίσης πιστεύω στο πολιτικό πλαίσιο η προενταξιακή βοήθεια, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και με τον ίδιο τρόπο, ο, όπως αναφέρονται και στην έκθεση της Επιτροπής, η όλη κατάσταση είναι νομικά δεσμευτική. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα του Κοινοβουλίου. Τρίτον, μετά από την βοήθεια του Κοινοβουλίου προβλέπονται κίνητρα στον κανονισμό, δηλαδή ε, οι χώρες ε, μπορούν να ανταμυφθούν ε, γιατί ενδεχομένως έχουν καταφέρει καλύτερα στο πλαίσιο της προνταξιακής βοήθειας. Τέταρτον, ο κανονισμός προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δείκτες έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν συμπεράσματα σχετικά με την βοήθεια που μπορεί να παρασχεθεί. Πέμπτον, το, τα κοινοβούλια κατόρθωσαν να διασφαλίσουν μέσα από κοινέ δηλώσεις τη χρηματοδότηση για μειονότητες και ε, όσον αφορά μάλλον όπως πρόκειται για όλους τους συμβιβασμούς, το Κοινοβούλιο πρέπει να δεχτεί κανονισμούς που προτείνει το Συμβούλιο και που αλλιώς εμείς δεν θα στηρίζαμε. Και εδώ αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στο θέμα των δικαιούχων. Πάντως, όπως σας είπα, στη συμβαστική πρόταση διασφαλίσαμε να ε, τηρηθούν οι προτεραιότητές μας και τελικά ο στόχος της διεύρυνσης να επεκταθεί και μετά το 2014. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας καλός συμβασμός. Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό για το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, τον κύριο Μάγια, τον κύριο Τάνοκ και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βιγγένιν, ο οποίος ε, πλέον ασχολείται με άλλα θέματα, με ε, διαφορετικά ε, προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι ο εισηγητής ο οποίος ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αποφασίσει το κορεπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων διδάχθηκα ότι όταν ο επικεφαλής ε, του Συμβουλίου λέει το κορεπέρ λέει όχι ε, τότε ήταν ε, όχι και όταν εγώ έκανα κάποιες προτάσεις το κορεπέρ έλεγε επίσης όχι. Οπότε έκλεινε το θέμα. Ωραία λοιπόν, θα δούμε κατά πώς το δικό μας κορεπέρ πει ναι. Λοιπόν, έχουμε μία ψήφο για το κάθε σημείο και γι' αυτό θα αναφέρω τις επιμέρους εκθέσεις και θα έρθω πρώτα, θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τους... Ε, ε, ποιος είναι υπέρ της έκθεσης. Abstimmung ist äh, Abstimmung ist jetzt. Ε, πέρας της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 0 κατά. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Τώρα θα ψηφίσουμε στην έκθεση... Όχι. Λάμπστορφ. Abstimmung ist geschlossen. της ψηφοφορίας. 44 προς Συγχαρητήρια κύριε Λάμστορφ, παρόλο που δεν είσαστε τόσο, πετύχατε τόσο πολλά όσο ο προηγούμενος Τώρα θα έρθουμε στο 6, ε, προταξιακή συνδρομή, ο κύριος ε, Ρούσεκ, του κυρίου Ρούσεκ, άρχεται η ψηφοφορία. Die Abstimmung ist 47 με 47 ψήφους υπέρ εγκρίνεται, δύο ψήφοι κατά, μηδέν αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν. Και τώρα θα έρθουμε στο εργαλείο γειτονίας του συναδέλφου Κουκράν. Άρχεται η ψηφοφορία. Die Abstimmung τη ψηφοφορία 46 προς 1 γίνεται δεκτή συγχαρητήρια. Εργαλείο γειτονίας, ε, εταιρική σχέση, συγγνώμη, Αντώνιο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 47 προς 0 εγκρίνεται. Δεν μου αρέσει αυτό το θετικό αποτέλεσμα, παρόλα αυτά συγχαρητήρια. Εργαλείο σταθερότητας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 47 προς 2 εγκρίνεται τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Μπιούτι Κόφερ και στην κυρία Μπραντνερ. Και τώρα συνεχίζουμε. Τώρα θα έρθουμε στην έκθεση για την Αλβανία. Ο κύριος Βούλιανιτς θέλει να μιλήσει, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους σκιώδεις εισηγητές και προς κάποιους άλλους από το, συναδέλφους από το Κοινοβούλιο που με βοήθησαν με τις συμβουλές που μου έδωσαν και τις υποδείξεις που μου έκαναν με σχέση με το πώς θα έπρεπε να προχωρήσω. Γιατί υπήρξαν κάποια εμπόδια. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Γραμματείας για την ευγένειά τους και το έργο τους. Ε, και ε, κυρίως για το γεγονός ότι ψηφίζουμε αυτό το ψήφισμα σήμερα. Εγώ άσκησα κάποια πίεση προσπαθώντας να γίνει, να διεξαχθεί η ψηφοφορία σήμερα και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια την προσεχή εβδομάδα. Από τη μία λόγω της κατάστασης της χώρας. Νομίζω ότι η χώρα μας το αξίζει. Και από την άλλη λόγω του Κοινοβουλίου, γιατί το Κοινοβούλιο πραγματικά αξίζει ε, να αποφανθεί ένα τέτοιο, για ένα τέτοιο θέμα πριν από την απόφαση του Συμβουλίου. Και πραγματικά πετύχαμε αρκετούς συμβιβασμούς και νομίζω ότι το ψήφισμα πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση και όλες οι τροπολογίες οι οποίες ε, κατατέθηκαν πηγαίνουν επίσης προς την ίδια κατεύθυνση ε, προσπαθώντας να αποδώσουν στην Αλβανία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Ε, παρόλο που εγώ συζητής ε, πέριψε ορισμένες από αυτές, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Ειλικρινά ελπίζω ότι θα εγκριθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και θα εγκριθεί επίσης από το Συμβούλιο ε, στα μέσα αυτού του μήνα. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους που με βοηθήσατε να κάνω αυτό το έργο γιατί πραγματικά δεν είχα τη σχετική εμπειρία ε, όταν έπρεπε να γίνει αυτή η εργασία αλλά νομίζω ότι όλοι μας πραγματικά έκαναν μια καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ και εγώ. Ε, συμφωνώ για το τελευταίο τμήμα των όσων είπατε, τουλάχιστον. Και θα ξεκινήσουμε τώρα την ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 1. Ποιος είναι υπέρ. Ε, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Στη συνέχεια για την τροπολογία 34 για το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα θα έρθουμε στην ε, τροπολογία... Eh, Βαστική τρία του κυρίου Σαλαφράνκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προτείνω μια προσθήκη σε αυτή την τροπολογία παριθμών 2 μέσω μια προφορική τροπολογία. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι πρόκειται για μια προφορική τροπολογία η οποία υπευλήθη από τον πρόεδρο τη Επιτροπή, ο οποίο είχε τοποθετηθεί ουδέτερα. Ήθελα να το κάνω εκ μέρου του ΕΛΚ για να χαιρετήσω την υπεύθυνη στάση τη ε, αντιπολίτευση σε αυτό το θέμα. Κύριος Ρούτσεκ, έχω ένα μικρό πρόβλημα με όλα αυτά. Δεν είμαι ε, κατά ως προς το περιεχόμενο, γιατί είναι σημαντικό στην, τόσο στην Αλβανία όσο και στις άλλες χώρες η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να συνεργαστούν. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα. Ε, και μακροπρόθεσμα. Αλλά έχω ένα πρόβλημα του διαδικαστικού ε, σε αυτή την, ε, όσον αφορά την ε, κατάθεση μιας προφορικής, υποβολή μιας προφορικής τροπολογίας σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μέσω της συνήθους διαδικασίας, γι' αυτό η ομάδα μου θα αντιταχθεί. Κύριε Ρούτσεκ, είναι κοινή τροπολογία μπορεί να γίνει κοινή τροπολογία εκ μέρους των σοσιαλιστών και του ΕΛΚ για την Ολομέλεια. Παρακαλώ. So we will oppose it now. Θα αντιταχθούμε αυτή τη στιγμή και θα δούμε, θα την καταψηφίσουμε και θα δούμε τι θα γίνει με την Ολομέλεια. Κύριε Σαλαφράγκα, κύριε... Πρόεδρε, ξέρουμε ότι επιτρέπει ο κανονισμός σε τέσσερα μέλη αυτής της ε, ε, Επιτροπή να αντιταχθεί σε μια προφορική τροπολογία. Είναι απλό το θέμα. Χθε όταν συζητήθηκε η έκθεση στην ομάδα μα, ομόφωνα ζητήσαμε αυτή η προσθήκη να συμπεριληφθεί, διότι είναι πάρα πολύ λογική. Κατανοώ ο κύριο Ρούσεκ και υποθέτω και οι τρεις άλλοι συνάδελφοι τον υποστηρίζουν. Το σημειώνω, σημειώνω τη στάση, ώστε το ΕΛΚ όταν η ομάδα του καταθέσει άλλες τροπολογίες να μπορέσουμε και εμείς να αντιταχθούμε. Πάντα η στάση μας ήταν ανοιχτή σε αυτή την Επιτροπή, ώστε να αποφασίζει ποιες τροπολογίες θα ψηφίσει και τις τροπορικές συμπεριλαμβανομένων η, η, ε, ολομέλεια μας. Α, Σαλαφράνκα, δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μιλάτε έτσι, κυρία Σαλαφράνκα θα πρέπει και εγώ στην ομάδα μου να τα συζητήσω αυτά τα πράγματα. Ελπίζω ότι με κατανοείτε. Όπως ελέγχθη λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε αντίθετοι ε, με την ψήφιση τους. Αλλά ας μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να βρούμε μια κοινή διατύπωση και να την ε, καταθέσουμε για να περάσει προς ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Αυτό ελπίζω ότι σας ικανοποιεί και επιτρέψτε μας και εμάς στην ομάδα μας να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε συζήτηση επί αυτού του θέματος. Συνεχίζουμε, λέει ο Πρόεδρος. Αρκετοί την καταψήφισαν, άρα δεν περνάει, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, προσπαθείτε να συνεργαστείτε και να παρουσιάσετε μία λύση για την Ολομέλεια. Αλλά θα σας πω το εξής. Το θέμα αυτό της Αλβανίας είναι θέμα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και πάντα ζητούσε η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση να να συνεργαστεί. Η παλιά κυβέρνηση οδήγησε σε μία ομαλή ε, μεταστροφή της κατάστασης και αλλαγή. Λοιπόν, και τώρα θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοια. Θα πρέπει όμως να το αναφέρουμε. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια η αντιπολίτευση δέχεται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό. Και τις δύο τελευταίες φορές δεν μπόρεσαν ούτε καν να προχωρήσουν και να καταλήξουν στο καθεστώς αυτός του υποψηφίου. Λοιπόν, καθυστέρησε η όλη διαδικασία, όπως ξέρετε, δύο φορές εξαιτίας αυτού του προβλήματος που υπήρχε μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα μιλώ ως μέλος του ΕΛΚ, όχι ως πρόεδρος. Έχω την εντύπωση ότι οι σοσιαλιστές, λοιπόν, ε, κάπως ε, κομματικά το παίρνουν το θέμα και όχι για το γενικότερο πολιτικό καλό. Λοιπόν, ας υπάρξει κάποια συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θετική λύση και πρόταση προς ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εντύπωσή σας είναι λανθασμένη, Πρόεδρε. Εγώ είπα ότι με την, ε, για την Αλβανία, για την Μακεδονία συνεργαστήκαμε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Διότι αν πρέπει να προσχωρήσουν οι χώρες αυτές και θέλουμε να προχωρήσουν, η, τα κυβερνώντα κόμματα και η αντιπολίτευση, όποιο κόμμα και να κυβερνά, πρέπει να συνεργαστούν. Τώρα, το ΕΛΚ ή κάποια άλλη ομάδα θα πρέπει να συνεργαστούν για να ευρεθεί λύση. Αυτή θα πρέπει να είναι η γραμμή πλεύσεως και νομίζω ότι εμείς από την ομάδα μας θα το κάνουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας προσπαθήσουμε να βρούμε μία συμβιβαστική διατύπωση για να προχωρήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε στην Ολομέλεια. Καταψηφίστηκε αυτή η προφολική τροπολογία, τελείωσε η συζήτηση. Δεν συνηθίζουμε εκ των υστέρων σε τέτοια θέματα να κάνουμε ε, ε, συζήτηση. Τα μέσα και τα εργασία τα συμβαστικά. Υπέρ, κατά... Πάμε στην τροπολογία 39, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 42, ε, όχι αυτή αποσύρθηκε, η 4 παρακαλώ, η σημαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 45 ε, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Ε, κάνουμε επαλήθευση. Έκλεισε η ψηφορία. Πάμε τώρα στην συμβαστική 5. Εγκρίνεται. Πάμε στην 47. Περ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 58 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην ε, τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 77 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 78 τροπολογία με προφορική τροπολογία υπέρ κατά υπέρ παρακαλώ κατά η τροπολογία ε, Κούκαν ε, γκρίθηκε. Η 64 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία Κορνέλισον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 η συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. εγκρίνεται 29 προς 22 ή 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι παρακαλώ υπέρ του πρώτου τμήματος, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ή 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος επαλήθευσης παρακαλώ για την 122. Εγκρίνεται. 28 23. Η συμβαστική 19 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 14. Συγγνώμη, τροπολογία 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 16 σε δύο τμήματα, υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται, υπέρ του δεύτερου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 30 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Για την 31 πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ, 3 υπέρ, 5 υπέρ εγκρίνεται, η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 και 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο της ε, πρότασης. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν. Θερμά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Κάνατε πολύ καλή δουλειά. Τώρα πάμε στην έκθεση Κατσίν. Ε, να ξεκινήσουμε κύριε Κατσίν με την ψηφοφορία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ευρύτατη πλειοψηφία και μπορούμε να μιλήσουμε ονομένοι όλοι. 14 τροπολογίες είναι τροπολογίες. Όχι, σε 40 τροπολογίες νομίζω ότι μπορέσαμε να έχουμε ε, ομόφωνη ε, άποψη υπέρ. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Είναι σήμερα εδώ ο κύριος Ντάτσι, ο Πρωθυπουργός και πάλι στην ε, ε Περισσότερες από 20 συναντήσεις έχουν γίνει σε ένα χρόνο. Πρόκειται για πραγματική ε, πραγματικό επίτευγμα των τελευταίων ετών. Έγιναν σωστά και οι εκλογές οι δημοτικές στο Κωσυφοπέδιο και χθε οι δημοτικές αρχές Κωσυφοπεδίου και Σερβίας συναντήθηκαν για πρώτη φορά εδώ και είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί τους. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται μόνο για υποστήριξη είναι ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα ότι πραγματικά μέχρι τώρα εκτιμούμε το ότι έχει διαδραματιστεί. Γι' αυτό θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να κάνω έκκληση και σε εσά και στην επόμενη γερμανική κυβέρνηση να κάνετε ό,τι μπορείτε για να μας βοηθήσετε να προχωρήσουμε περαιτέρω αυτό το Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Η κυβέρνησή μου θα κάνετε και η δική σας κυβέρνηση ε, προσπαθεί να κάνει. Πιστέψτε με. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πάντα να ταυτοποιούμε μόνο μία κυβέρνηση. Ε, το καλό πρέπει να λέγεται για όλους. Καμιά φορά όταν γίνεται κανένα κακό πάντα ένας είναι αυτός τον οποίο ψέγουμε. Αλλά ας σταματήσουμε να ενεργούμε έτσι. Äh, λοιπόν, ε, ξεκινάμε με τη συμβαστική 1, γιατί η, τροπολογία 10 αποσύρθηκε. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 2 συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 26 τροπολογία υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 37 υπέρ, μισό λεπτό, 37 παρακαλώ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 52 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκε. Κοιτάξτε, στην ψηφορία συμμετείχε έτσι κι αλλιώς το ΕΛΚ που απέριψε. Όλοι οι άλλοι ψήφισαν υπέρ. αυτό έκλεισε ψηφοφορία και αυτή τη φορά ε, δικαιώθηκε το ΕΛΚ, το ECR δεν είχε συμμετάσχει. Παρακαλώ όμως να συμμετέχετε στην ψηφορία τουλάχιστον ο συντονιστής της ε, πολιτικής ομάδας, ακόμα και αν αυτό είναι κοπιαστικό. Η 53, ε, η 55 τώρα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Charles, είναι δυνατόν, σας παρακαλώ, κάποιος από την ομάδα σας να συμμετέχει ε, στην ψηφοφορία, γιατί στην τελευταία ψηφοφορία κανείς δεν σηκώσε το χέρι του ούτε υπέρ ούτε κατά ούτε τίποτα. Ε, νοερά ίσως να συμμετέχετε αλλά ε, δεν συμμετέχετε ε, σηκώντας το χέρι. Και να κάνουμε συνεχώς ηλεκτρονικές ψηφοφορίες αυτό κοστίζει. Γιατί εσείς λέτε συνέχεια να εξοικονομούμε χρήματα αλλά δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία. Λοιπόν, πάμε στη συμβιβαστική 64. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 υπέρ κατά αποχές, 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Λοιπόν, εγκρίνεται η τροπολογία η 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τον επιμένει κανείς και αυτό είναι μία μέτωση. Λοιπόν, η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 85 τροπολογία υπέρ κατά ξαναψηφίζουμε παρακαλώ είναι όχι η 85 η 85 εγκρίθηκε 86 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ 93 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 96 υπέρ, κατά ε, εγκρίνεται. Η 99 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ Η 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλλον εγκρίνεται. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 22-25. Πάμε στην 136. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 όχι, 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Οι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, υπέρ γιατί είναι τις ε, κατά αποχές απορρίπτεται, Οι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 2 και 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο, παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε τώρα στην τροπολογία για το κοσυφοπέδιο. Ε, ποιος την αντικαθιστά παρακαλώ, γιατί δεν είναι παρούσα η κυρία Λούνατσεκ. ή 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την 15. Πάμε στην 19 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Κοίταξε, Μπέντσε, παρακαλώ πες στους ανθρώπους σου από την ECR να συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Κάνω τάρτη τώρα, Εγκρίνεται. Η συμβαστική 1, υπέρ κατά εγκρίνεται. Πάμε στην 31 τροπολογία, παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές, για την 34 παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για την 63 παρακαλώ υπέρ κατά Το ECR, οι συντηρητικοί μεταρρυθμιστές, είναι υπέρ, υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 73 υπέρ το, του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ του δεύτερου τμήματος κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 70 παρακαλώ τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 74 σε δύο τμήματα. Υπέρ του πρώτου τμήματος παρακαλώ. Κατά ε, αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Äh, äh, äh, der Antrag είναι angenommen. Εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 76. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση. Στην Die Abstimmung ist geschlossen. Und πέρας της ψηφοφορίας 31 ε, ε, προς 14 γίνεται δεκτή. 105 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπερθμών 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 6 δύο τμήματα υπέρ, για το πρώτο τμήμα, ε, κατά εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, 11 ε, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ε, Πασέσκου Πρέντα και Μίλαν Μον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με μικρή πλειοψηφία ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. 39 ναι, 3 όχι, 4 αποχές. Θερμά συγχαρητήρια. Τώρα θα έρθουμε στην έκθεση αυτή που έχει πολλές ελπίδες για το μέλλον. Η έκθεση Πρέντα για την Ισλανδία. Κύριε Πρέντα, θέλετε να πείτε κάτι. Τότε θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμών 3. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. 44 ναι, 0 όχι, 0 αποχές, θερμά συγχαρητήρια. Τώρα θα έρθουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης, την έκθεση Γκόμες. Εν, Άννα. Θα ξεκινήσουμε με το 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, δεν πρόσεξα, λέει ο πρόεδρος, ποιος είναι υπέρ του 32. Κατά, κατά, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 χωριστή ψηφοφορία, τμήμα 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 έχει καταπέσει. 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ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 κατά, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, ποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Abstimmung ist geschlossen. 31 ja, 3 nein, 8 Enthaltungen. Ένα, ναι, 8 όχι, 3 αποχές. Συγχαρητήρια Άννα. Τώρα θα έρθουμε στην έκθεση προόδου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Äh, Πρέπει εδώ να κάνουμε γρήγορα ούτως ώστε ε, να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα. Στις 11-12 ε, του είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, γιατί σήμερα έχουμε τον εκπρόσωπο της Αλβανίας εδώ. Στις 11.30 θα πρέπει μέχρι, τώρα, ε, μέχρι τότε να έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση αυτής της έκθεσης. Η συνάδελφος κυρία Πάκ έχει το λόγο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, σκέφτηκα ότι εκ, να υποβληθεί η έκθεση την οποία είχαμε υποβάλει το Μάιο να υποβληθεί και πάλι, γιατί τελικά δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στη Βοσνία Ριζεγοβίνη αλλά δεν φταίνε οι άνθρωποι, αλλά ένα σύνταγμα το οποίο συντάχθηκε σε μια στρατιωτική βάση στο Οχάιο και το οποίο δεν πληρεί τις προποθέσεις ενός δημοκρατικού κράτους. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε η απόφαση του Δικαστήριου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, για την υπόθεση Σέντζι Φίτσι ε, που λέει ότι ο καθένας θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα ε, για την Προεδρία και μόνο οι Άζας δεν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα. Αυτό είναι αδύνατον σε ένα δημοκρατικό καθεστώς. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει κάτι το οποίο εσφαλμένα έχουν συντάξει κάποιοι άλλοι άνωθεν. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση. Ε, καταρχήν, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εάν δεν γίνει αλλαγή, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτέ εκλογέ το επόμενο έτο. Γι' αυτό το λόγο ο κύριο Φούλε διαπραγματεύθηκε 16 ώρε με την πολιτική ηγεσία τη χώρα χωρί να καταλήξουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Στη χώρα αυτή έχουμε και άλλα πολύ σημαντικά προβλήματα που έγκυται στο ότι σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και βεβαίως μεταξύ των διαφόρων εφροντήτων, συγγνώμη. Και γι' αυτό η κατάσταση επιτοπίως είναι πολύ δεινή. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, για παράδειγμα, όπου δεν είναι να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Υπάρχουν ε, ε, αδιέξοδα ε, όσον αφορά πολλές δικαστικές ε, αποφάσεις ε, που δεν εφαρμόζονται, άλλες που εκκρεμούν. Είπα ότι έχουμε δύο θέματα. Από τη μία έχουμε δύο ντότες, την Κροατική Βοσνιακή Ομοσπονδία, η οποία επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα γιατί τους έχει υπαγορευτεί το καθεστώς στην Ουάσιγκτον. Έχουμε δέκα καντόνια έχουμε περίπου 150 υπουργού οι οποίοι προσπαθούν ένας να βάλει τρικλοποδιά στον άλλον. Δηλαδή έχουμε τις τοπικές, τους τοπικούς φορείς, από πάνω έχουμε τα καντόνια και έχουμε και μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει και από πάνω Υπάρχει και η βοσνιακή ε, κυβέρνηση. Ζητούμε λοιπόν, απαιτούμε από τους ανθρώπους να μπορούν ε, να ενεργήσουν σε μια κατάσταση όπου αυτό είναι αδύνατον. Το πρόβλημα ωστόσο δεν έγκυται στην αλλαγή αυτής της λειτουργίας αλλά ε, στο γεγονό ότι οι αλλαγέ των θεσμικών οργάνων δεν μπορούν να γίνουν από εμά, πρέπει να γίνουν από τους ίδιους. αν υπάρχουν 11 για παράδειγμα υπουργοί παιδεία σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατό για να γίνει αποδεκτό έστω και ένα πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ούτως ώστε να εφαρμοστεί ο δικό ε, χάρτη ε, υψηλού επίπεδου ε, και να υπάρξει μια σταθερότητα. Η Βοσνία Ζεγοβίνη είναι πολύ πίσω, είναι προτελευταία και στη συνέχεια ε, και τελευταίο το Κόσοβο. Ε, θα πρέπει οι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι θα, εμείς εργαζόμαστε για το δικό τους συμφέρον. Το πρόβλημα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης είναι επίσης η γενικευμένη διαφθορά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του επιχειρηματικούς κύκλους και τους πολιτικά ηθήνοντες που πραγματικά διαδραματίζουν, ε, μια, πραγματικά αποτελούν μάλλον μια πολύ δυσάρεστη συντροφιά. Και ε, ελπίζω πάρα πολύ να υπάρξει μια αλλαγή, αλλά δεν μπορούμε να απευθύνουμε μια έκκληση και να την διατυπώσουμε ρητά. Ίσως αυτό βοηθήσει να ξεσηκωθεί ο πληθυσμός και να πούν στους πολιτικούς τους τελεία και παύλα μέχρι εδώ. Δεν υπάρχει ε, ε, υποστήριξη εκ μέρου των πολιτικών για μεταρρυθμίσει που όμω είναι αναγκαίε. Χρειάζονται μεταρρυθμίσει στο εργατικό δίκαιο, χρειάζονται μεταρρυθμίσει όσον αφορά τις, ε, την εσωτερική διάρθρωση, αλλά ακόμα και την ιατρική πολιτική. Εδώ και δέκα τουλάχιστον χρόνια απαιτούμε επιτέλους στον τομέα αυτό να γίνει κάτι, ούτως ώστε προϊόντα της γεωργικής πολιτικής να, από τη γεωρική παραγωγή συγγνώμη, να μπορούν να εξάγονται. Αλλά πάντοτε ε, ακόμα όλα αυτά δεν έχουν λυθεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει η καλή πρόθεση εκ μέρους πολιτικής ηγεσίας. Και το άσχημο είναι ότι δεν είναι ε, τα ε, θεσμικά όργανα που παρεμποδίζουν αυτές τις εξελίξεις, αλλά ηγέτες των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι ε, δεν έχουν κανένα πολιτικό αξίωμα εντός αυτών των οργάνων και παρόλα αυτά το κάνουν. θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε την πολιτική ηγεσία. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τίποτα άλλο και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους συγκετεύσουμε να κάνουν κάτι. Έχουμε τα ΙΠΑ, τα ταμεία ΙΠΑ, τα οποία δεν, ε, ε, δεν αξιοποιούνται γιατί δεν υπάρχει συμφωνία σε σχέση με το ποιο θα πρέπει να αποφεληθεί από αυτά τα κονδύλια. Άρα υπάρχει τεράστια καταστασία σε όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι είναι λογικό εκ μέρου τη Επιτροπή να σκεφτεί κατά πόσο ε, πρέπει να δοθούν αυτά τα κονδύλια από αυτά τα ταμεία, τα IPA, IPA για διευκρινίζοντας ποιοι θα επωφεληθούν, ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα και επιπροσθέτως υπάρχει το πρόβλημα από την δεκαετία του 90 ότι έχουμε πάρα πολλούς ε, πρόσφυγες που επιθυμούν να επιστρέψουν, να επαναπατριστούν. Πολλοί το έπραξαν, αλλά όχι όλοι. Και γι' αυτό θα πρέπει να ε, επισημάνουμε αυτό το πρόβλημα. Για παράδειγμα, ε, στα βόρεια της Ρεπουμπλίκ Σέρψκα, ε, δεν τον φέρω ρητά, αλλά αυτή την περιοχή εννοώ, η οποία πραγματικά από την εποχή του πολέμου έχει απολύτως καταρρεύσει. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως αγροτική οικονομία. Ε, παλαιότερα ήταν ε, ε τόπος για κατάσταση κρατικών βιομηχανιών. Ε, πάρα πολλοί λοιπόν επιθυμούν να επιστρέψουν. Κάποιοι επέστρεψαν, έφτιαξαν σπίτια, αλλά δεν έχουν ούτε νερό, ούτε ρεύμα, ούτε απολύτω τίποτα. Ε, δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι δυνατόν να φτιάχνουν σπίτια οι άνθρωποι και τελικά να αποκλείονται από την κοινότητα γιατί δεν έχουν καμία πρόσβαση στις ε, ε, κοινή ωφέλεια. Ε, δεν μπορώ παρά λοιπόν να απευθύνω μια έκκληξη να γίνει κάτι στον τομέα αυτό. Και υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν έχω αναφέρει ρητά στην έκθεσή μου. Για παράδειγμα μια περιβαλλοντική πολιτική όπου θα μπορούσαν να τεθούν ενδεχομένω κάποια θέματα. Ε, κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Δεν ε, συνέταξα αυτή την έκθεση για να ψηφιστεί με τις άλλες εκθέσεις, γιατί πάντοτε παραμένω με την ελπίδα ότι θα μπορέσω να πω επιτέλους κάτι ε, θετικό, ότι 16 ώρες που πέρασε ο Φιούλε με τους, πολιτικά, με τους πολιτικούς ηγέτες, τελικά θα καταλήξουν κάπου, θα καρποφορήσουν ε, και να εφαρμοστεί η απόφαση Σέτζνικ ε, Φίντσι. Και αυτή η προπόθεση για άλλα προβλήματα θα πρέπει να επιληθούν και στον τομέα της παιδείας, ε, της ε, ε, προσχολικής, της φύλαξης των παιδιών κλπ. Λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω τίποτα θετικό. Ελπίζω οι πολιτικοί πριν από τα Χριστούγεννα να μπορέσουν να καταλήξουν σε, μια, σε κάποια ολοκλήρωση, σε κάποιο τέλος, σε κάποια έκβαση, ούτως ώστε επιτέλους να μπορέσει να εφαρμοστεί το σύμφωνο σταθερότητας. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις, για αυτή την πολύ καλή παρουσίαση του θεσμικού διεξόδου στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, αλλά και επίση αυτό το οποίο αναφέρθηκε στην έλλειψη βούληση εκ μέρου των πολιτικών προκειμένου να επιτευχθεί μια αλλαγή εκεί. Για την... Η κυρία Γκόμες έχει το λόγο. Όχι, ο κύριος Ρούτσεκ. Σήμερα κυρία Μποσκότσι δεν μπορεί να είναι εδώ και εξ ονόματό της θα πω το εξή. Χαιρετίζει την έκθεση της κυρίας Πακ διότι θα μπορέσει για την όλη διαδικασία της προσχώρησης Βοσνία ε, να αποτελέσει μία κάποια πρόοδο. Κάτι προσβεύει τον Οκτώβριο του 2014, όπω ελέγχθη όμω δεν υπάρχει ε, καμία ουσιαστική ε, όλο το θεσμικό θέμα είναι πολύπλοκο, δεν υπάρχουν ακόμη συμβιβασμοί και οι διάφοροι ηγέτες δεν διευκολύνουν την καθημερινή ζωή του πολίτη και δεν ε, υπάρχει πρόοδος. Επίσης πρέπει να προσθέσω ότι υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας και αυτό είναι κάτι το οποίο φύγει ιδιαίτερα στους πολίτες και το μέλλον. Στο κυρία Μποσκό θα ήθελε να υπάρχει καρποφόρο συνεργασία με την κυρία Πάκ. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να αποδείξουμε στους πολίτες της Βοσνίας ότι δεν εγκαταλείπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χώρα της, αλλά όπως είπε και η Ντόρις οι πολιτικοί ηγέτες, οι ηγέτες των πολιτικών κομμάτων είναι αυτοί που έχουν ε, τη μοίρα της χώρας αυτή στα χέρια τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρούτσεκ. Η κυρία Λέντσε εξονόματης της Άλντε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εκ μέρους των ε, σκιωδών εισηγητών και του συναδέλφου να πω κάτι. Δεν έχω να προσθέσω ε, πολλά μετά από την εξαιρετική παρουσία της Doris Πακ. Δυστυχώς αυτά που ε, ελέγχθησαν είναι η πραγματικότητα. Η σκληρή πραγματικότητα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να υποδείξω είναι να προσθέσουμε μια έκκληση, να κάνουμε μια έκκληση στην ε, επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να κάνει μία από τις πρώτες προτεραιότητές της το θέμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης διότι με μεγάλη ενεργητικότητα και χωρίς μεγάλες ευκολίες προχωρήσαμε τώρα στα θέματα της Σερβίας και του Κοσφοπεδίου και το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση αυτή διότι χωρίς μεγάλη δέσμευση δεν μπορεί κανείς να αναμένει πρόοδο για τον λαό της Βογνίας Ερσεγοβίνης. Βεβαίως όλοι θα πρέπει να θέλουν να συμμετάσχουν δυναμικά και θετικά σε μια τέτοιου είδου άσκηση αν πρέπει να αρχίσει δηλαδή συνεργασίες και βελτίωσης εάν το επιθυμούν όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πάκ, την εισηγήτρια. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι εξαιρετικά απογοητευτικά αυτά που ακούσαμε, διότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή τη απόφασης Edgic Φίντσι είναι πρωταρχική σημασία και θα πρέπει να γίνει ένα κάπως και οργανωμένο κράτος η Βοσνία ριζεγοβινη Δεδομένου ότι δεν έχουμε προς το παρόν κανένα αποτέλεσμα, καμία πρόοδο, θα πρέπει να μην ε, κατεβάσουμε τα χέρια, αλλά να περιμένουμε κάτι να γίνει. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η Ανεμή Νίτς προηγουμένως. Ότι δεν θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να του εγκαταλείψει. Είναι πρωταρχικής όμως σημασίας να συνεχίσουμε ε, ενωμένοι όσον αφορά την ε, ε, σχέση μας και την πρόοδο που θέλουμε να επιτευχθεί στην Βοσνία Ερζεγοβίνη από μία φωνή και με την διεθνή κοινότητα. Θα καταθέσουμε τροπολογίες και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε κάπως να βελτιώσουμε αυτή την πολύ καλή έκθεση, αλλά με τόσα πολλά προβλήματα. Για... Ο κύριος Τάνο και ο κύριος Βουλιάνιτς, ποιος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. διότι έχει κατανοήσει μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση πώς έχει πώς έχουν τα πράγματα στη Βοσνία Ζεγοβίνη και η κυρία Πακ έχει πιάσει το νόημα. Υπάρχουν πολλά υποσχόμενες και θετικές προοπτικές σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, στη Βοσνία Ερσεγοβίνη, αλλά τα πάντα είναι στατικά αυτή την εποχή. Εδώ και αιώνες έχουν μάθει να συνυπάρχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τρεις διαφορετικές θρησκείες, τρία-τέσσερις έθνη αν θέλατε, αποκαλούνται σεράια, κοινοί άνθρωποι. Αυτοί που δεν ξέρουν πώς να συνεπάρχουν βεβαίως είναι οι πολιτικοί στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η συμφωνία του Ντέιτον ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να σταματήσει ο πόλεμος. Σταμάτησε ο πόλεμος. Αλλά δεν υπάρχει μηχανισμός για να οργανωθεί αυτή η χώρα. Και δεν μπορεί κανείς να οργανώσει μια χώρα ε, βασιζόμενος μόνο σε ειρηνευτικές συμφωνίες. Είναι απόλυτα σαφές ότι τουλάχιστον συγκεκριμένη περίπτωση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης αυτό το σύστημα δεν λειτουργήσε. Αυτή τη στιγμή γίνονται στο Σαράγεβο διάφοροι επαιτειακοί εορτασμοί για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ευρώπη έχει αναλάβει να κάνει κάτι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι πολιτικοί εκεί δεν έχουν μάθει να κάνουν συμβιβασμούς. Γιατί κανένας δεν τους υποχρέωσε ποτέ. Δεν υποχρεώσει θυκάνουν και έτσι απαντούν στα πάντα με τα όπλα. Δεν έχουν μάθει τίποτα. Θα πρέπει όμως να το μάθουν. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να τους υποχρεώσουμε να μάθουν πώς να κάνουν συμβιβασμούς. Η πολιτική πίεση δεν είναι ωραία λέξη. Δεν είναι δημοκρατικός όρος, αλλά θα πρέπει να τον εφαρμόσουμε εδώ και βεβαίως έχει απόλυτη σχέση με το χρήμα που θα πέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε να κάνουμε με μικροσερίφιδες σε τοπικό επίπεδο. Uh, και ο καθένας θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα της εθνότητάς του. Θα πρέπει όμως η Βοσνία Ερζεγοβίνη να κάνει βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η έκθεση, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να ασκεί περισσότερη πίεση προς τους πολιτικούς της Βοσνίας Ερσεγοβίνης, καθώς και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να οργανώσουν την ε, απαραίτητη αυτή πίεση για να υπάρξει πρόοδος. Ο κύριος Πόσελτ. Äh, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να πω το εξή. Τέθη το ερώτημα κατά πόσον από την τελευταία έκθεση για τη Βοσνία προέκυψαν θετικέ εξελίξει, Όχι, έγινε κάτι θετικό. Το τι, εντωμεταξύ η Κροατία είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον σύνορα με τη Βοσνία Ερτζεγοβίνη. Αυτό ε, δημιουργεί βέβαια προβλήματα, αυτό το γνωρίζουμε, θέματα ηθαγένεια και πολλά άλλα. Από την άλλη πλευρά βέβαια, είναι και μία μοναδική ευκαιρία να υπάρξει διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την άμεση ε, γειτονία, δηλαδή συνεργασία με τις ε, παραμεθόριες περιοχές έτσι ώστε και αυτές να ευδοκιμήσουν και να μην διοχετεύονται όλα τα κονδύλια μέσω Σαράγεβο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η Βοσνία Ερσεγοβίνη έχει πλέον σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τώρα, όσον αφορά στο Σύνταγμα, έχει απόλυτα δίκιο η κυρία Πάκ και τη είμαι ευγνώμων που το λέει με αυτή τη σαφήνεια που το λέει. Δηλαδή, ε, οι, τα Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερικής, όχι εμεί, επιβάλλαν, επέβαλαν το Σύνταγμα στην Βοσνία Σεγοβίνη. Τέλειωσε τότε ο πόλεμος, καλό αυτό. Όμως ε, αυτό το Σύνταγμα δεν προωθεί την ειρήνη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν το Σύνταγμα. Και ε, πρέπει να πω ότι σε αυτή τους την προσπάθεια δεν πρέπει να του εγκαταλείψουμε. Μάκροπρόθεσμα υπάρχουν δύο ε, κίνητρα και δύο οι οποίοι παράγοντες που είναι πολύ σημαντικοί είναι αυτοί οι νέοι που είτε φεύγουν είτε κατεβαίνουν στους δρόμους. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την πολιτική παιδεία, τους νέους, να βοηθήσουμε να εκπαιδευτεί μια νέα γενιά πολιτικών. Και πρέπει να ε, στηρίξουμε και την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί νομίζω ότι η χώρα μπορεί να εννοηθεί μόνο από κάτω. Η ε, πολιτική παιδεία, η υποστήριξη των νέων και η τοπική αυτοδιοίκηση αυτοδιοίκηση. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ. Κάποιος ίσως από τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση, ε, να λάβει το λόγο. Πολλές φορές έχει υπογραμμιστεί ότι θέλει και η Ευρωπαϊκή πτυχή, γενικότερα η κοινότητα, την ε, Βοσνία να ε, προχωρήσει και η εκτέλεση της απόφασης Σέτζικ Φίντζι είναι ένα πρώτο βήμα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ε, Βόσνιους να δημιουργήσουμε γέφυρες για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Αυτό είναι δικό μας καθήκον. Είναι προτεραιότητα λοιπόν και νομίζω ότι ο Επίτροπος δεν θα είχε περάσει 16 ώρες χωρίς να σταματήσει και χωρίς να κοιμηθεί αν δεν ήταν προτεραιότητα για αυτό το θέμα. Και αμέσως μετά έστειλε και πάλι μία ομάδα στην Βοσνία και συνεχίζονται συζητήσεις για να μπορέσουν να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να πω ότι όλα τα θέματα τέθηκαν επί τάπητος, κάποια θέματα ε, λύθηκαν αλλά δεν μπορέσαμε να ε, καταλήξουμε σε τελική συμφωνία, διότι δεν μιλάμε για τελική συμφωνία αν δεν επιληθούν όλα τα επιμέρους προβλήματα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την ε, απόφαση, την Selgic Finchi και αν δεν λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, μιλήσουμε για ολοκλήρωση συμφωνίας. Όταν λοιπόν αυτή η απόφαση ολοκληρωθεί και φτάσουμε σε απόφαση, θα ζητήσουμε το Φεβρουάριο του Υπουργού να προχωρήσουν. Αλλά εάν δεν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την συμφωνία και παραμείνουν παραμείνει η κατάσταση όσο έχει και πρόκειται για μια παγιωμένη κατάσταση που δεν προχωρεί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και βεβαίως Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Και ξέρουμε ότι οι πολίτες επέδειξαν ενδιαφέρον και έχουν ασκήσει και μεγάλη πίεση στους ηγέτες τους για να μην ε, καταρακώσουν όλες τις προσπάθειες και τις προοπτικές της προσέγγισης της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5 Μαΐου είναι η μέρα στην οποία θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ε, συνταγματικές αλλαγές που προβλέπονται και οι τροποποιήσεις ώστε να δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεως και να ισχύσουν για τον επόμενο Οκτώβριο που θα γίνουν εκλογές με το νέο Σύνταγμα. Ξέρουμε ότι ο χρόνος παίζει εναντίον μας και πρέπει όλες αυτές οι συμφωνίες να επιτευχθούν ώστε να γίνουν οι εκλογές τους τον επόμενο χρόνο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, όπως είπε και η συγγεντρία, αν ε, δεν γίνουν σωστά τα πράγματα ε, και δεν μπορέσουμε να σεβαστούμε τις ημερομηνίες και να πετύχουμε συμφωνία, θα ε, έχουμε αρνητικές επιπτώσεις για τις επόμενες εκλογές. Και για την όλη διαδικασία ευχαριστώ. συντομία θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Η κυρία Νάιτς είπε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε οι άνθρωποι εκεί να κατανοήσουν ότι εμείς πραγματικά παίρνουμε σοβαρά τα, όσα, αιτήματά τους. Ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει πολλοί επικεφαλής ε, ηγέτες κυβερνήσεων ε, οι ενότατε εξωματούχοι να μεταβούν εκεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. Ναι, μεν πήγε ο κύριος Σέρνσεν, ο ύπατος εκπρόσωπος επίσης, ο οποίος ε, προσπαθεί να κάνει κάτι. Αλλά αν φτάσει κάποιος με ένα πολύ γνωστό πρόσωπο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν για παράδειγμα πήγαινε εκεί η καγκελάριος Μέρκελ και έκανε εκεί μια ομιλία έτσι όπως και στον Βελιγράδι, ίσως ορισμένοι πραγματικά θα διαπίστωναν ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται για αυτούς και ίσως θα άλλαζαν και τη συμπεριφορά τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσουμε τις κυβερνήσεις όχι μόνο το 2014 να μνημονεύουν την έναρξη του πολέμου, ε, αλλά τελικά να συμβάλλουν ε, ενεργά ε, προς την ειρήνευση. Και νομίζω θα πρέπει να το διατυπώσω αυτό και ρητά. Σας ευχαριστώ και πάλι και είμαι πρόθυμη να καταθέσω και κάποιες άλλες τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολύ, Ντόρι. Στις 11 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. στι 6 το απόγευμα. Και με αυτό ολοκληρώνουμε. Περνούμε στο επόμενο, η Σαουδική Αραβία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος στην Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική. Πρόκειται για πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεση, Θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Αναγκόμες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή των συναδέλφων στο γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη έκθεση που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Σαουδική Αραβία. Τουλάχιστον από όσων μπόρεξα να δω εγώ, επισκέφθηκα την Σαουδική Αραβία πριν από τρεις εβδομάδες για να συλλέξω πληροφορίες ο κύριος Μάρτσιν από την γραμματεία μας με συνόδευσε, καθώς και ένας πάλι ο κύριος Μαμαντόφ. Κάναμε μία πολύ καλή επίσκεψη σε επίπεδο ανωτάτου επίπεδου κυβερνητικού. Μας διευκόλυναν επίσης για να συναντήσουμε και ε, εκπροσώπους της ε, ε, πολιτικής κοινωνίας. Ο πρέσβης επίσης μας βοήθησε και με συνόδευε και ένα, μια νέα κυρία, νέο μέλος της Σούρα, όπως ξέρετε 13 γυναίκες, 30 γυναίκες πλέον είναι οι νέες εκπρόσωποι της ε, ε, διαβουλευτικής συνέλευσης, έχουν συμβουλευτικό ρόλο στην Σούρα. Πρόκειται για μια χώρα που είναι πολύ σημαντική για μας. Από κάθε άποψη, εμπορική, οικονομική, και σημαντικός εταίρος για την περιοχή παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα, ερωτηματικά και αμφιβολίες. Πρόκειται όμως για σημαντικό εταίρο για την περιοχή και για τον κόσμο. Έχουμε βεβαίως να κάνει μια χώρα που δεν έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Έχει μια μοναρχία η Σούρα ε, έχει περιορισμένες εξουσίες η, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει ότι η ανεξιθρησκεία είναι εγγυημένη και ο καθένας μπορεί να ασκεί τα θρησκευτικά του ε, δικαιώματα στους δικούς του λατρευτικούς χώρους, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, υπάρχει σκληρό Ισλάμ έχουμε να κάνουμε με το λίκνο του Ισλάμ. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό βεβαίως δεν αποτελεί δικαιολογία και δεν ε, συνάδει με τις υποχρεώσεις ε, της Σαουδικής Αραβίας βάσει των συμβάσεων που έχει υπογράψει. Ένα άλλο πρόβλημα οφείλεται στο γεγονός και αυτό μπορέσαμε να το διαπιστώσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις εξαιτία του γεγονότες ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ ιδιάζουσα χώρα. Έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ συντηρητικό Ισλάμ, με τους Χαμπίς, οι οποίοι είναι τους Βαχαμπίς, οι οποίοι είναι πάρα πολύ, ε, είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν την κατάσταση, συμπεριλαμβαμένες κυβέρνηση και της βασιλικής οικογένειας και η ερμηνεία του Ισλάμ όντως αποτρέπει τη χώρα από το να ανοίξει, να αναπτυχθεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε σε συνεδριάσεις και με μέλη της κυβέρνησης και με την βασιλική οικογένεια. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη ένταση και στην πράξη τι είδαμε. Παρά το γεγονός, είδαμε τι συμβαίνει με την κατάσταση των γυναικών. Παρά το γεγονός ότι την δεκαετία του 50 του 60 ασκήθηκαν πολύ μεγάλες πιέσεις εκ μέρους των ΙΠΑ ώστε να έχουν ε, την δυνατότητα να σπουδάσουν τα κορίτσια. Και έτσι σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία πάρα πολλές μορφωμένες γυναίκες που αγωνίζονται για την πράσιση των δικαιωμάτων τους σε πολύ σκληρές συνθήκες και γι' αυτό έχετε στην Σουρά αυτές τις 30 πολύ ικανές γυναίκες και σε διάφορες άλλες ε, θέσεις διαπραγματευτών και ε, στην ε, κυβέρνηση υπάρχουν τρομερές διακρίσεις. Επισκεφτήκαμε πανεπιστήμιο την πριγκίπισσα Νόρα Υπάρχουν υποδομές, αν θέλετε, για τις γυναίκες, αλλά είναι κάπως απομονωμένες κάπου. Αλλά είναι παρούσες, προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην κοινωνία και θέλουν να έχουν ε, πρόσβαση σε θέσεις στο λιανικό εμπόριο φεριπίν Φερρυπίν θα θέλανε να μπορούν να ε, πολλούν εσόρουχα. Πώς είναι δυνατόν να πουλούν οι άντρες εσόρουχα για γυναίκες σε αυτή τη χώρα αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε να κάνουμε όντως με διακρίσεις, μπόρεσαν ε, με την επιμονή τους ε, να κατακτήσουν ε, αυτό το είδος των εμπορίων και τώρα κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσουν να εμπλακούν σε άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Ε, από τους ε, πανεπιστημιακούς φοιτητές και από τους διπλωματούχους το 60% είναι γυναίκες, είναι πολύ μορφωμένες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει μεγάλη διαφορά στην κοινωνία αυτή σε χρόνια και σήμερα αρχίζει και φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά την άδεια οδήγησης, ξέρετε τι δημιουργήθηκε πριν από ε, λίγο καιρό και τι δημοσιότητα δόθηκε. Υπουργό των φάνηκε να είναι υπέρ τη χορήγης άδεια οδήγηση της γυναίκας, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοια. Κάνουν ό,τι μπορούν. Είπανε ναι, αλλά καμία δεν έχει άδεια οδήγηση, άρα δεν μπορεί να οδηγήσει. Και υπάρχει ένα σύστημα μεσαιωνικό κυδαιμονία των γυναικών, αν θέλετε. Κάποιος πάντα κυδαιμονεύει μια γυναίκα ο πατέρα, ο αδελφός, την ε, συνοδεύει παντού, ο άντρας της, εν πάση περιπτώσει. Ένα αρσενικό πάντα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μου το είπαν πάρα πολλές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων και γυναικών μελών της ε, βασιλικής οικογένειας, αλλά μας είπαν κάποιες άλλες, ακούστε, είναι για τη δική σας προστασία. Σαν να φοράτε ζώνη προστασίας υποχρεωτικά στο αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και λίγοι υπεφωτισμένοι σε αυτήν την κοινωνία μεταξύ των ανδρών. Αλλά κάποιοι μου εξήγησαν ε, ως παραδοσιακές αξίες κάποια θέματα που θεωρούμε εμείς προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελεύθερη άσκησή τους. Βεβαίως δεν υπάρχουν καμήλες στους δρόμους. Πρόκειται για μια σύγχρονη κοινωνία. Έχουμε να κάνουμε με εργατικούς και ικανούς ανθρώπους και με εντυπωσίασαν πάρα πολύ πολλά μέλη κοινωνίες. Υπάρχουν όμως και προβλήματα μειονοτήτων με τους ΙΤΕΣ, με τους ε, ε, μετανάστες εργαζόμενους επίσης υπάρχει πρόβλημα. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες εργαζόμενοι. Περίπου 9 εκατομμύρια λοδαποί ζουν στην Σαουδική Αραβία, οι περισσότεροι είναι μετανάστες. Υπάρχει όπως καταλαβαίνετε το θέμα της ασφάλειας, όπως και εδώ, ακόμη πιο οξύ στην Σαουδική Αραβία, διότι πολλοί φοβούνται ότι διεισδύουν ε, τρομοκράτες και συστήνουν τρομοκρατικές οργανώσεις από, τις, από άλλες χώρες. Και μου είπαν ότι υπάρχει το πρόβλημα της σαουδικοαραβοποίησης, αν μου επιτρέπετε αυτή την αδόκιμη λέξη. Τι σημαίνει αυτό, ότι όσο περισσότερο κανείς έχει πρόσβαση σε παιδί, όσο περισσότερο μορφωμένος είναι, τόσο περισσότερο θέλει να δεχτεί στην κοινωνία και το πρόβλημα είναι ότι οι θέλουν όλες τις ε, εργασίες, τις ωραίες, να τις κάνουν οι μορφωμένοι οι Σαουδάραβες, αλλά ποιος θα είναι ο ρακοσυλέκτης ή ο δοκαθαριστής, κάποιος ο οποίος δεν έχει εξειδικευτεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες από την Αιθιοπία, αλλά και από άλλες χώρες. Υπάρχουν ε, περίπου... Ε, 8.000 χιλιάδες οι οποίες φτάνουν με 12 πτήσεις καμιά φορά την ημέρα. Υπάρχουν όμως πάντα προβλήματα, ε, ε, υπήρξαν σειράξεις, ε, τρεις ε, θάνατοι και οι μεν επιρρύπτουν το λάθος τους δε. Εμείς πήγαμε σε μία ενδιαφέρουσα περίοδο όταν έγινε η αναγγελία των ε, συζητήσεων που θα γίνονταν σε ανώτατο επίπεδο για τα πυρηνικά όπλα με το Ιράν. Υπάρχει μεγάλος ε, ανταγωνισμός μεταξύ των δύο κρατών αυτών και δεν είναι μόνο το πρόβλημα, ε, διαφορετικών ε, θρησκευτικών ακραίων ε, θέσεων. Ξέρουμε ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ήδη από τη δεκαετία του 70 μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας για θρησκευτικού λόγους και όταν πήγαινα στην Σαουδική Αραβία διάβαζα διάφορα άρθρα από διάφοροι υψηλού επίπεδου μέλη της οικογένειας της ε, βασιλικής που έλεγαν ότι αισθάνονται κάπως προδομένοι από τους Αμερικανούς γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχε αρνηθεί σε επίπεδο ο ΙΕ ε, την θέση ενός μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας στην Σαουδική Ερεβία και μετά από την ε, εξαιρετικά ε, δυναμική ε, εκστρατεία την οποία είχαν κάνει, αισθάνθηκαν ότι είναι προδομένοι από τους Αμερικανούς και θέλησαν να σηκωθούν να φύγουν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το θέμα της Συρίας. Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει την συμμαχία κατά του Ασάντ. Καλό είναι αυτό, αλλά και έχει και αρνητικές ε, επιπτώσεις, διότι προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ισχυρός οικονομικός ε, παράγοντας και ελέγχει όλες τις χρηματοπιστωτικές ε, ε, συναλλαγές που γίνονται σε όλη την ε, περιοχή η Σαουδική Αραβία. Υπενθυμίζω την 9η ε, Σεπτεμβρίου και βεβαίως η Σαουδική Αραβία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα των τρομοκρατικών επιθέσεων και ότι αυτό σημαίνει τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως δεν μπορούν να ελέγξουν τα ποσά τα οποία διακινούνται στα πλαίσια ε, ε, ε, φύσεως αν θέλετε φιλανθρωπικών ε, έργων τα οποία χρηματοδοτούνται. Επίσης, το θέμα της αποκατάστασης των πρώην φυλακισμένων του Αγουαντάναμο έχει ε, σημασία στη χώρα αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιθέσεις λοιπόν. Στη Συρία είδαμε ότι υπάρχει και ανταγωνισμός. Και δεν μπορούσαν να μας εξηγήσουν γιατί υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός μεταξύ Κατάρ και Σαουδικής Αραφίας με υποστήριξη εκ μέρους κάποιων, ε, κάποιων τρομοκρατικών ομάδων. Αυτό όμως δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει Οι Αμερικανοί αποφάσισαν ε, ε, τελικά να μην επέμπουν στη Συρία. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μετά από την, ε, τις αντιδράσεις, από, πριν της απογοήτευση και διαβάσαμε κάποια άρθρα τα οποία προσυπογράφουν μάλιστα και σημαντικά μέλη της βασιλικής οικογένειας σε σχέση με την Τουρκία και λένε ίσως ε, αν δεν υπάρχει το Ιράν, να καταφύγουμε στο Πακιστάν για την ε, πυρηνική του ομπρέλα, που στη τελική ανάλυση του χρηματοδοτήσαμε κιόλα. Ξέρω ότι αυτή δεν είναι βέβαια η επίσημη γραμμή και έχετε πάρει και όλοι σα ε, κάποια ενδιαφέροντα σχόλια από την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας που Αυτά όλα είναι κάποια περίληψη, μπορούμε αν θέλετε να τα εμπλουτίσουμε. Αυτό που θέλω να πω, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία και παρατηρήσεις που έκανε ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με αυτά τα σχόλια είναι σχόλια του πρέσβη πολύ πιο πρόσφατα, πιο θετικά ε, σχετικά με την ε, πυρηνική συμφωνία με το Ιράκ Μία νέα λοιπόν σχέση προκύπτει πλέον με το Ιράν. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχα πάει στο Ιράν και οι Ιρανοί είχαν δείξει κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό δεν αποκλείεται και νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Θα χρειαζόμουν πάρα πολύ χρόνο για να επεκταθώ. Φαντάζομαι δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα όμως να σας επισημάνω κάτι. Να σας επισημάνω το εξής ότι η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών θα επεκταθεί. Είχε προβλεφτεί μέχρι τις 10, αλλά επειδή θα ψηφίσουμε τέλη Ιανουαρίου, θα έλεγα η προθεσμία να πάει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου. Έτσι ώστε οι συνάδελφοι να δουν και τα σχόλια των Σανταράβων και την έκθεση με την ησυχία τους να καταθέσουν τροπολογίες οι οποίες ε, πραγματικά θα εμπλουτίσουν την έκθεση. Και κάτι πριν κλείσω. Κοιτάξτε, η έκθεση αυτή δεν αφορά την ε, Σαουδική Αραβία, ε, αφορά ε, και γενικότερα το ρόλο της Βόρειας Αφρικής και των χωρών με Αραβική Άνοιξη. Υπάρχουν αντιφάσκουσες απόψεις. Στην Λιβύη ο μουφτής είπε ότι δεν είναι καλό να οδηγούν οι γυναίκες. Αυτό βέβαια το είχε πει και ένας ιερέας στη Σαουδική Αραβία. Όμως στη Σαουδική Αραβία μου είπαν όλοι ότι αυτόν τον αγνοούν όλοι. Δεν θεωρείται κάποιος που να επηρεάζει καταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Έχει όμως σημασία να δείξουμε πώς αυτός που τον περιφρονούν οι Σαουδάραβες τον εκμεταλλεύονται άλλοι που αναφέρονται στη Σαουδική Αραβία, αναφέρομαι προφανώς ε, στην ιδιαίτερα συντηρητική πτέρυγα του Ισλάμ, το εκμεταλλεύονται λοιπόν για να διαδώσουν πολύ δυσάρεστες και αρνητικές απόψεις σε χώρες όπως είναι η Λιβύη, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του ε, να οδηγούν οι γυναίκες ή όχι και άλλα, ότι οι δασκάλες θα πρέπει να καλύπτουν το πρόσωπό τους ας πούμε. Ίσως αυτή να μην είναι η επίσημη πολιτική της Σαουδικής Αραβίας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ε, ακραίοι στη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι ε, δίνουν τροφή να ξεσηκωθούν και άλλοι ακραίοι στη δική μας τη γειτονιά. Σας ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννάκο από το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Γκόμες για την έκθεση που εξεπώνησε η πραγματικότητα είναι προφανής. Πρόκειται για ένα καθεστώς ε, θρησκευτικού φονταμενταλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται από την υψηλή ηγεσία η οποία ταυτόχρονα λόγω των οικονομικών μέσων που διαθέτει απολαμβάνει όλα τα αγαθά της δύση όταν εξέρχεται στη Δύση και διαβιώνει όπως διαβιώνουν στη Δύση. Απ' την άλλη πλευρά το οικονομικό πλαίσιο της χώρας για τους πολλούς είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή το μέσο κατακεφαλήν εισόδημα σε σχέση με τα συνολικά εισοδήματα της χώρας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και βέβαια είναι εξευτελιστικά χαμηλή η μισθή των ε, τριτοκοσμικών που έρχονται στο, στη Σαουδική Αραβία να δουλέψουν και ζουν κάτω από πολύ δυσάρεστες συνθήκες. Όχι μόνο εκεί, αλλά και ε, στα Εμμυράτα. Θα γνωρίζετε ίσως το προπέρσινο γεγονός εδώ στις Βρυξέλλες όταν α, πριγκίπισσα των, της Σαουδικής Αραβίας κατέπλευσε στο ξενοδοχείο Κόνρατ με 20 δούλες εκ των οποίων μία μίλησε στο ξενοδοχείο και επενέβη ο εισαγγελέα. Τα ίδια έγιναν ακριβώς από μία αντίστοιχη κυρία στις Ηνωμένε Πολιτείες στη Φλόριντα. Δεν είναι λοιπόν μόνο τι γίνεται εκεί μέσα, αλλά είναι ότι περιφέρονται ανά τον κόσμο με τα συστήματα αυτά και είναι λυπηρό. Η θεωρία που αναπτύσσεται εκεί είναι ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν σιγά σιγά, ότι μια φορά στα δέκα χρόνια μπορεί να αφήνουν και καμία γυναίκα να οδηγήσει αυτοκίνητο και άλλα τέτοια επίσης ότι κάποιες γυναίκες μπορεί να έχουν ένα δίπλωμα νομικής αλλά τι νομική υπεράσπιση να κάνουν ε, όταν η Σαρία έχει κατακυρωθεί ε, με βάση τα δυσμενέστερα στοιχεία για τους πολίτες. Σας υπενθυμίζω την περσινή υπόθεση μιας μικρής κοπέλας από τη Ζιλάνκα που εκτελέστηκε γιατί τη θεώρησε υπεύθυνη η μητέρα του παιδιού όταν πέθανε το παιδί της, ένα μωρό. Και παρά τις προσπάθειες των δυτικών και όλων δεν κατέστη δυνατόν να γίνει απολύτως τίποτα. Ε, η υπόθεση αυτή κύριε Πρόεδρε είναι προφανής και έρχεται και σε σύγκρουση με αυτά που λέμε εμείς και βάζουμε ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θυμάστε την ταλαιπωρία που είχαμε για να κλείσουμε την ιστορία του Καναδά. Ζητούσαμε από τον Καναδά να, να δεχθεί μία ρήτρα για ανθρώπινα δικαιώματα και εδώ τώρα ποιε είναι οι σχέσεις μας με όλους αυτούς. Δηλαδή ποιος πιστεύει ότι θα εισακουστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε οτιδήποτε. Εδώ το καθεστώς αυτό ξεκινά από το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι περίπου ζώα, δηλαδή ο μισός πληθυσμό. και από εκεί και πέρα και ότι ο υπόλοιπο λαός είναι έτσι, διότι το χρήμα όλο συγκεντρώνεται στη βασιλική οικογένεια. Επομένως, τι να πει κανείς. Βεβαίως θα υπάρξουν τριβές, έχουν ζητήσει να μας δουν οι πρέσβεις και όλα αυτά. Α, ισχυρίζονται ότι αυτό είναι θέμα θρησκείας. Αλλά αν η θρησκεία είναι πολιτικό σύστημα, τότε τι είδους συνομιλητές μπορεί να έχει στην Ευρώπη ένα τέτοιο σύστημα. Και επομένως κύριε Πρόεδρε έχω την αίσθηση ότι θα καταλήξουμε να γίνει μια έκθεση η οποία θα είναι σχετικά προσεκτική στις διατυπώσεις. Υποθέτω εκεί θα καταλήξουμε. Αλλά κανείς από εμά δεν πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει η χώρα αυτή και τα συστήματα αυτά τα οποία αναπτύσσονται και μάλιστα και εις βάρος θρησκευτικών αποκλήσεων του Ισλαμισμού ότι θα μπορέσουν ποτέ να λειτουργήσουν υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διότι είναι δομημένα έτσι γιατί έτσι συμφέρει. Και επομένως, τι να σας πω κύριε Πρόεδρε, να κλείσει η Ευρώπη τις πόρτες σε όλους αυτούς. Είναι πάρα πολύ δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολλές οι χώρες και η επιρροή που έχει ασκηθεί από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία στην Αφρική είναι πολύ δυσάρεστη. Ε, εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγαινα στο σχολείο δεν μαθαίναμε τι είδου θρήσκευμα υπάρχει στο, στην Αφρική. Μπορεί και να θεωρούσαμε ότι επρόκειτο για ειδωλολατρικές προσεγγίσεις και τέτοια. Και τώρα ξαφνικά έχουμε μάθει ότι είναι όλοι μουσουλμάνοι, φονταμεταλιστές, συγκροτούν τρομοκρατικές ομάδες κτλ. Και ποιοι πληρώνουν τους τρομοκράτες, αυτά είναι ερωτηματικά που όλοι ξέρουμε τις απαντήσεις. Βεβαίως οι χώρες αυτές δεν έχουν πια τόση σημασία για το ενεργειακό όσοι είχαν στο παρελθόν. Όταν η Ευρώπη ξυπνούσε και κοιμόταν με το φόβο των τιμών του πετρελαίου που θα αποφασίσει ο ΟΠΕΚ στη Βιέννη. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να εκφράσουμε όλη τη δυσαρέσκειά μας για την κατάσταση αυτή. Διότι η Σαουδική Αραβία είναι προφανές ότι την τροφοδοτεί σε όλο τον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει και αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη στην εξωτερική της πολιτική δεν έχει κάποιον ισχυρό λόγο. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας και αυτά που συνέβησαν τώρα με την Κορανία και την Αρμενία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε ακόμη δεν έχει καταλάβει κανείς μας πώς με τόσο ενθουσιασμό είδαν την Αραβική Άνοιξη. Γιατί είδατε τα πράγματα που κατέληξαν. Επομένως είναι απογοητευτική η κατάσταση. Φλιβερή. είναι εναντίον του ανθρωπίνου κεφαλαίου και πρέπει να βρεθούν τρόποι οι χώρες αυτές να πιεστούν ισχυρότερα, να λάβουν το μήνυμα ότι πρέπει να κάνουν κινήσεις συγκεκριμένες που να αποδεικνύουν ότι σέβονται στοιχειοδός τον άνθρωπο. Τώρα για την θανατική ποινή θα σας πω ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσω της Σαρία ερμηνεύουν το Κοράνι όπως θέλουν. Δηλαδή μου εξηγούσε κάποιος ότι μπορεί να πεις ότι σε καταδικάζω σε θάνατο, αλλά μπορεί να πεις και σε συγχωρώ. Αλλά αυτοί διαλέγουν να καταδικάζουν σε θάνατο, να κόβουν χέρια και άλλα τέτοια, τα οποία είναι επικώς ανατριχιαστικά. Και καταλαβαίνω κύριε Πρόεδρε την, το ενδιαφέρον και τα συμφέροντα και της Ένωσης γιατί αποτελεί υποτίθεται ένα πυλώνα σταθερότητας στη Σαουδική Αραβία. Εγώ θα βάζα πολλά ερωτηματικά και σε αυτό και ας αφήσουμε την κυρία Κόμες, να συνεννοηθούμε και όλοι μαζί, να φτιάξουμε κάτι μέσο που να μην ενοχλεί και τόσο πολύ που θα μας κλείσουν, που θα, που θα τους κάνει να να γίνουν τελείως αρνητικοί αλλά να στέλνει και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Είναι από τα αδιέξοδα κύριε Πρόεδρε. Είναι από τις αδιέξοδες καταστάσεις. Γιατί έχουν τους ενεργειακούς πόρους και γι' αυτό τα κάνουν αυτά. Και επομένως εγώ δεν θα ήμουν ευτυχής να έχω φιλίες με τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, ε, ε, Μαριέτα. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο. Η κυρία Νεμινίτς από την Άλντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ την Άννα για το κουράγιο και την αποφασιστικότητά της να αναλάβει ένα θέμα που είναι πολύ δύσκολο και εξαιρετικά λεπτό. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό με συνεκτικό τρόπο αυτό είναι κάτι το οποίο μας το εξήγησε και η κυρία Γιαννάκου στην ε, παρέμβασή της. Το πρόβλημα το πραγματικό είναι πραγματικά τι είδους σχέσεις μπορούμε να αναπτύξουμε με χώρες σαν την Σαουδική Αραβία γνωρίζοντας πώς έχει εσωτερική κατάσταση της χώρας. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενθαρρύνουμε αλλαγές διότι είναι σαφές ότι άλλαξαν κάποια πράγματα, βεβαίως με αργούς ρυθμούς. Επίσης είναι σαφές και θα έπρεπε να είναι σαφές ότι η παρούσα κατάσταση ίσως παρά τη, αυτά τα οποία είπε η προηγούμενη συνάδελφος να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι πάντα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι πιο ε, ριζοσπάστης από σένα και να εκφράζει ριζοσπαστικές ιδέες. Και για να μπορέσουμε να ε, εισαγάγουμε μερισσότερη περισσότερη ελευθερία σε τέτοιου είδους κοινωνίες όπως η Σαουδική Αραβία, γιατί αυτή είναι δημοκρατικά Απ' την άλλη μπορείτε να έχετε επιτάσεις των αντιθέτων φαινομένων, περισσότερη τρομοκρατία και σκληροπυρηνικούς. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι θα πρέπει να είστε περισσότερο αυστηρός ε, και να σφίγγετε περισσότερο τα λουριά. Είναι δύσκολος λοιπόν αυτός ο δρόμος που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Αλλά όπως είπε και η Άννα, και εγώ επίσης σε, ε, στο παρελθόν πολλές φορές επισκέφθηκα με διάφορες αντιπροσωπείες την Σαουδική αραφία Συζήτησα εγώ με γυναίκες μορφωμένες του επιστημονικού κόσμου πολιτικές. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το επίπεδο και υπάρχουν Πολλοί οποίοι υποστηρίζουν τον προσανατολισμό τον σωστό και τις εξελίξεις στην ε, Σαουδική Αραβία. Αλλά νομίζω ότι και εμείς και όλοι και ίσως περισσότερο από τις είπα χρειαζόμαστε το πετρέλαιο που παράγει η χώρα αυτή. Το να διακόψουμε σχέσεις εξαιτία της δινής κατάστασης των ανθρωπίων δικαιωμάτων δεν είναι εναλλακτική λύση, θα ήταν πολύ αρνητικό. Ας είμαστε ε, πραγματικά ειλικρινείς και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι και σωστό για την ισορροπία των γεωπολιτικών θέσεων. Όντως, οι μουσουλμανικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από πηγές ε, της περιοχής όλο και περισσότερο διεισδύουν και στην Αφρική. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα πρέπει να το λάβουμε όπως αλλά από την άλλη γιατί τους αφήνουμε πεδίο δράσης. Γιατί τους δίδουμε τέτοιου είδους δυνατότητες να ενεργήσουμε τον τρόπο αυτό. Με την Άννα Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έγιναν για να συντάξουμε μία έκθεση ισοσκελισμένη. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόχμπιλ, παρακαλώ ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ακόμη ένα θέμα να συζητήσουμε πριν να έλθει ο πρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας, γι' αυτό να είμαστε παρακαλώ όσο πιο σύντομοι γίνεται. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Άννα Γκόμες για αυτή την πολύ καλή έκθεση και οι δικές μας συστάσεις, οι τροπολογίες θα έλεγα, σχετίζονται κυρίως με, την, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω ότι μπορούμε να εξετάσουμε το καθεστώς αυτή τη στιγμή της Σαουδικής Αραβίας στην ε, Γενέβη ε, όπου γίνεται μια σωστή εξολόγηση με τα, με τις, ε, των μεταρρυθμίσεων και των ελλείψεων όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Εγώ έχω κάποιες τροπολογίες που ίσως βοηθούν σε μια ακριβέστερη διατύπωση όταν αναφέρεστε στην κατάργηση της θανατικής ποινή, εμείς θα θέλαμε να καταθέσουμε μια τροπολογία λέγοντας ότι ενθαρρύνουμε μια περαιτέρω μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος ώστε να καταργηθούν όλες οι μορφές σωματικής ε, ποινή. Τώρα, όλοι οι παράγραφοι που αναφέρονται στα, στις μη κυβερνητικού οργανισμούς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ έχουμε καταθέσει σχετικά κάποιες τροπολογίες γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να μπορούν να εργάζονται κανονικά, νομίμως να έχουν το δικαίωμα να αναπτύσσουν εκεί τις δραστηριότητές τους. Επίσης, τροπολογίες σε σχέση με αυτό το οποίο εξαγγέλθηκε κατά τη διάρκεια της δικής μου επίσκεψης πριν από δύο εβδομάδες ότι μελλοντικά θα είναι πιο εύκολο για τους διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επισκέφτονται τις φυλακές και τα κρατητήρια και επίσης να παρακολουθούν ε, δίκες, διεξαγωγή δικών. Ε, θέματα σημαντικά ε, και που αφορούν τη μοίρα των αντιφρονούντων. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση των μεταναστών εργαζόμενων εκεί, και εδώ έχουμε καταθέσει κάποιες σχετικές τροπολογίες, σημειώνοντας επίσης ότι τον ε, Ιούλιο έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις ε, σε σχέση ε, βελτιώνοντας τις σχέσεις εργαζόμενων και εργοδοσίας. Ε, τώρα, όσον αφορά αυτό το σύστημα των ανδρών συνοδών και ε, ανδρικής κυδαιμονίας των γυναικών και το θέμα της εκπαίδευση εκπαίδευσης ανωτά του επίπεδου για τις γυναίκες. Έχουμε καταθέσει και εδώ κάποιες σχετικές τροπολογίες. Ε, επίσης, όσον αφορά την αναγνώριση του Συμβουλίου ΣΟΥΡΑ και των κανονικών θεσμικών σχέσεων με το δικό μας κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε καταθέσει μια τροπολογία τονίζοντας την σημασία ε, κοινωνικής δεκτύωσης μέσω του διαδικτύου. Αυτές είναι οι πρώτες ε, Αυτές είναι οι τροπολογίες μας και Άννα είπε στην προφορική σου παρουσίαση ότι θέλεις να ζητήσεις από την κυβέρνηση να υποστηρίξει και τις εξελίξεις στο Ιράν, ιδιαίτερα τη συμφωνία όσον αφορά τα πυρηνικά. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι αυτό είναι σαφώς ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και θα ήθελα να καλέσω και τους πράσινους συναδέλφους και την ε, Άννα ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν και τα ίδια κριτήρια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αντιμετώπιση των γυναικών τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στο Ιράν αλλά αυτή η έκθεση δεν αφορά αποκλειστικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι ξεκάθαρο για μένα ότι το βασίλειο της Αδικής Αραβίας έχει ένα πολύ ε, εντόνως κατασταλτικό σύστημα ιδιαίτερα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, των μη ε, μουσουλμάνων κλπ. Αλλά η έκθεση αυτή παρουσιάζει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, άρα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάτω από την προοπτική της εξωτερικής πολιτικής το βασίλειο της Αδικής Αραβίας υπήρξε σύμμαχος της Δύσης κατά της Ιρανικής, ε, ε, του Ιρανικού επεκτατισμού ε, σε σχέση με το θέμα του Ιράκ και των κρατών του κόλπου. Και η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας σε αντίθεση με το Ισραήλ έγινε ευπρόσδεκτη στη Γενέβη ε, όσον αφορά, σε σχέση με το πάντα με το θέμα του πυρηνικού, ε, με το θέμα του εμπλουτισμού του Ιρανίου στο Ιράν. Τώρα, όσον αφορά την υποστήριξη του Κατάρ ε, για αυτές τις ομάδες, πραγματικές ομάδες της Τζιχάντ, υπάρχουν αποδείξεις για άμεση υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, της Αλκαΐντας στο Μάλι γιατί η κυβέρνηση το αρνείται και λέει ότι υποστηρίζουν μόνο το Εθνικό Συμβούλιο της Συρίας. Αλλά προφανώς υπάρχουν κάποιες ατομικές πηγές που, λειτουργούν, που δίνουν ανεξάρτητα, χρήματα ανεξάρτητα από τις κυβερνητικές πηγές το ίδιο το Βασίλειο και ο Ιμπν Σαούντ έχουν υποστεί επιθέσεις από την Αλκαΐντα. Άρα η κατάσταση είναι κάπως εγκεχημένη και εγώ συμφωνώ ότι οι ομάδες σαλαφιστών διασυνδέονται με την Αλκαΐντα, το Ισλαμικό Μακρέπ, την Αλσαμπάπ κλπ. Όλες αυτές τις εξτρεμιστικές, φονταμεταλιστικές, ισλαμιστικές ομάδες που δρούν στην Αφρική, στη Βόρεια Αφρική. Βεβαίως ε, και υπήρξε ένα πρόγραμμα εκ μέρους των Wahhabi χρηματοδότηση στην Αιθιοπία αλλά και χώρες της Δυτικής Βαλκανικής όπως είναι η Μακεδονία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη ε, που μας, ε, πράγματα που μας ανησύχησαν γιατί υπήρξε μια ριζοσπαστικοποίηση της αλβανικής κοινότητας στη Μακεδονία και υπήρξε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου εν σχέση με φαινόμενα εθνικού και θρησκευτικού εξτρεμισμού. Και επίσης όσον αφορά το 16 και το 19 για το Zero Sum Game. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η διατύπωση και θα ήθελα να καταθέσω κάποιες τροπολογίες εκ μέρους του CCR ούτως ώστε να μετριαστεί κάπως η γλωσσική διατύπωση της έκθεσης και να στηρίξουμε κάπως, να χαιρετήσουμε το γεγονό ότι ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας έκανε κάποια βήματα στο χώρο της εκπαίδευσης, παραδείγματα που γυναίκες ε, μπορούν να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω τι εννοεί η Άννα με αυτό το zero-sum game. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Και τώρα θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στον πρέσβη της ε, Σαουδικής Αραβίας για να ακούσουμε και τις δικές του σκέψεις. Αλλά κύριε πρέσβη, ε, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μιλήσετε πολύ δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες ε, και τους άλλους συναδέλφους Ελπίζω η επίσκεψη που έκανε στη χώρα μου να τους ικανοποίησε. Θα είμαι σύντομος γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και σε τελική ανάλυση δεν είναι και δική μου δουλειά να πω στα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το τι πρέπει να κάνω. Απλά εγώ θέλω να παραθέσω κάποια στοιχεία για όλους. Εγώ είμαι εδώ για να σας αποδείξω ότι η κυβέρνησή μου η της Σαουδικής Αραβίας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη και με ιδιαίτερο σεμβασμό τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και να διασφαλίσουμε ότι η σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σαουδική Αραβία ε, θα είναι επίσης όρης πάντα και θα μας οδηγήσει και προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να διαβεβαιώσω την κυρία Αναγκόμες ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Ε, δεν υπάρχουν πια σε εμάς μεσαιωνικοί νόμοι και διατάξεις. Και αναφέροντας και τέτοιου είδου χαρακτηρισμούς, νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει. Θέλω επίσης να διαβεβαιώσω όλους ότι η Σαουδική Αραβία ήταν και εξακολουθεί να είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας και την ευημερία ε, σε όλους τους εταίρους δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για το ρόλο της ε, Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα ή το εμπόριο. Τα τελευταία 20 χρόνια η ευρωπαϊκές εταιρείες χρονια οι ευρωπαικες συνάψει συνάψεις ε, ε, με τη Σαουδική Αραβία που ισούνται με 800 δις μέχρι και ένα 3 εκατομμύρια δολάρια. Για να κλείσω κύριε Πρόεδρε, Εμείς ε, είμαστε μια χώρα που στρέφει το βλέμμα προς το μέλλον με αισιοδοξία. Ξέρουμε ότι το μέλλον της χώρας μας είναι στα χέρια των νέων. Η παιδεία, παιδεία και πάλι παιδεία αυτή είναι η σωστή λύση που πρέπει να προαχθεί. Και αυτό κάνουμε εμείς. Πριν από 55 χρόνια οι γυναίκες δεν πήγαιναν στο σχολείο, επίσημα τουλάχιστον. Τώρα έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο γυναίκες, μάλλον, 1,5 ε, εκατομμύριο φοιτητές. Το 52% είναι γυναίκες. Έχουμε περίπου 600.000 φοιτητές ε, και επίσης και σε αυτά τα πανεπιστήμια το 54% είναι γυναίκες. Έχουμε 160.000 φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και το 35% εξ αυτών είναι γυναίκες. Έχουμε ε, δικηγόρους, ε, κατόχους διδακτορικών ε, διατριβών. Πρόσφατα η Guardian δημοσίευσε αυτά τα στοιχεία. Και αν είχα περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου, με μεγάλη μου χαρά να σας υπέβαλα και άλλες στοιχεία. Μπορούμε να ανητούμε και κατηδίαν και να σας αποδείξω ότι στη χώρα μου έχουν λάβει χώρα πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Πραγματικά δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας και αν έχει την καλοσύνη η Άννα μόνο για ένα λεπτό γιατί πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες για την ε, ε συνεισφορά τους, κυρίως τον κύριο Πρέσβη για να έχουμε περαιτέρω συζητήσεις, πάντα το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ότι συζητώντας περιβέρω μπορούμε να κατανοήσουμε μεν τους 10 καλύτερα και αμοιβέ να επηρεάσουμε και την κατάσταση. Εμείς πραγματικά, όπως ξέρετε, θέλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβουμε δεσμένες για να προχωρήσουν τα πράγματα. Και εντάξει, η διατύπωση ίσως κάποιες φορές είναι ατυχής, τώρα αυτό με το μεσαιωνικό. Εγώ απλώ προσπάθησα να περιγράψω κάτι σε σχέση με τις διεθνείς δεσμεύσεις. Και βεβαίως θα πρέπει το θέμα των οικονομικών σχέσεων και γενικότερα των σχέσεων με εμάς να επικεντρώσει την προσοχή μας. Χρειαζόμαστε περισσότερο ε, χρόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε την ε, σωστή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι, λέει ο Πρόεδρος, Ζήτησα την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών ως τις 6 Ιανουαρίου, λέει η κυρία Γκόμες, διορθώνοντας τον Προεδρεύοντα. Θα ψηφίσουμε τέλος Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου, άρα θα πρέπει να έχουμε χρόνο. Θα έχουμε χρόνο. Εντάξει, θα το συζητήσουμε αργότερα. Ακούστε, προς το παρόν αναφέρεται 10 Δεκεμβρίου, αλλά θα το συζητήσουμε. Το επόμενο θέμα είναι ο περιφερειακός ρόλος του Πακιστάν και οι πολιτικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπόρις Ζάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο, γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Το Πακιστάν ε, ίσως μας παρουσιάζεται σαν μια απομακρυσμένη χώρα, παρόλα αυτά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή και ε, ταυτόχρονα είναι ένα σημαντικό παίκτη στο διεθνές στερέωμα. Καταρχήν όσον αφορά την δημόσια μάχη κατά τη δημόσια, κα, ε, παγκόσμια μάχη κατά της τρομοκρατίας καθώς και τις σχέσεις με την ε, Ινδία που είναι αρκετά πολύπλοκες, καθώς και το ρόλο του Πακιστάν στο Αφγανιστάν μετά την απόσυρση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά, όλα αυτά είναι κάποιες ε, προϋποθέσεις που τονίζουν τη σημασία του ρόλου του Πακιστάν και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να πάρει μια ξεκάθαρη στάση το δεύτερο κομμάτι αφορά τις εξελίξεις εντός του Πακιστάν, τα εθνικά ζητήματα και πρόκειται εδώ για μια διαδικασία η οποία προσωμιάζει με την ε, πραγματικότητα της Σαουδικής Αραβίας και για να το πούμε κάπως απλουστευμένα ε, ε, πρόκειται εδώ για θεοδερχικού τύπου ε, σχέσεις και φαινόμενα στο Πακιστάν όπου βεβαίως παρόλα αυτά έχουμε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και η πρώτη δημοκρατική ε, μετάβαση έλαβε χώρα στο Πακιστάν και Βεβαίω είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τι δημοκρατικέ δυνάμει στο Πακιστάν. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Στο Πακιστάν υπάρχουν μεγάλε περιοχέ οι οποίες δεν υπάγονται στην ε, εξουσία του κράτους. Και ε, το κράτος ε, δεν είναι ενοποιημένο υπό την κλασική έννοια ε, υπάρχει, υπάρχουν οι διάφορες ε, φυλές και υπάρχουν περιοχές που ελέγχονται από φυλές. Ε, γι' αυτό είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Πακιστάν. Το πιο σημαντικό κομμάτι βεβαίως είναι η διαπραγματεύση με τους Ταλιμπάν και εδώ το ζητούμενο είναι να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχουμε εμείς οι ίδιοι ε, με τους Ταλιμπάν στη δική μας χώρα και ε, από την άλλη τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, στη γειτονική χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να επιληθούν όλα αυτά για να σταθεροποιηθεί η ειρηνευτική διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα το ζητούμενο είναι ο εκδημοκρατισμός της χώρας ούτως ώστε να, οι κανόνες του παιχνιδιού να ε, γίνουν δημοκρατικοί. Είναι σημαντικό βεβαίως για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο να μειωθούν οι εντάσεις στην περιοχή. Από τη μία θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις συνομιλίες με τους Ταλιμπάν, από την άλλη ε, δεν θα πρέπει να προδώσουμε τις δημοκρατικές μας αρχές. Αυτό είναι το δίλημα ενώπιον του οποίου βρισκόμαστε. Και υπάρχουν στρατηγικά προβλήματα σε δύο επίπεδα. Από τη μία η συνεργασία με τη ΣΥΠΑ, γιατί στην περιοχή είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμόζει μια ανεξάρτητη πολιτική ως πραγματικός εταίρος των ΙΠΑ στην ε, περιοχή αυτή. Και μια τελευταία παρατήρηση. Και σε αυτή την έκθεση είχαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ε, της ε, λεγόμενης ε, στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Αυτή είναι μια έννοια η οποία θα πρέπει να οριστεί ακριβέστερα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σαν ένα ουσιαστικό εργαλείο άσκησης πολιτικής γιατί από μια ρεαλιστική οπτική γωνία η έννοια αυτή της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ε, είναι κάτι μη ρεαλιστικό όσον αφορά τουλάχιστον την πραγματικότητα του Πακιστάν. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να οριστεί εκ νέου. Uh, uh, of the is uh, Πολύ Ζάλα. Ε, έρθει ο εκπρόσωπος, ο, ο πρόεδρος του Αλβανικού Κοινοβουλίου. Θα δώσει το λόγο στον κύριο Γκάλερ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο γιατί σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με αυτά που μας είπε. Και επίσης ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδουμε σε αυτή τη σημασία την, σε αυτή τη χώρα τη σημασία που της προσήκει. Η χώρα έχει προβλήματα, έχει το Αφγανιστάν γείτονες, την Ινδία. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να βοηθήσουμε στη χώρα αυτή και νομίζω ότι υπάρχουν τρία θέματα που είναι σημαντικά και όπου πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Η αναπτυξιακή συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτής ε, θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι ώστε οι νέοι να έχουν καλή παιδεία και να μην καταλήγουν σε αυτά τα μαντράς, ε, τα θρησκευτικά σχολεία, ε, τα οποία σίγουρα δεν είναι προσαρμοσμένα στον 21ο αιώνα. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα οικονομικά. Έχουμε το GSP συν. Ε, αυτό πρέπει να το επικυρώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Και νομίζω αυτό είναι σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και όσον αφορά την προαγωγή της δημοκρατίας, ε, να μην κάνουμε μόνο παρακολούθηση εκλογών. Εγώ έχω πάει ε, τώρα, είχαμε το 2008, αλλά και τώρα έχουμε τη συνέχεια αυτών των προγραμμάτων και εργαζόμεθα ουσιαστικά για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Γι' αυτό λοιπόν στο σημείο 13 η διατύπωση που έχει επιλεγεί δεν είναι και πάρα πολύ σωστή, διότι κατά την άποψή μου, ε, εδώ είμαστε σαφείς, στα αγγλικά λέει, ε, θεωρεί ε, την δημοκρατική εκπαίδευση στο Πακιστάν ότι θα πρέπει να ακολουθεί μια πιο ξεκάθαρη στάση όσον αφορά την παροχή βοήθειας. Κοιτάξτε, Όλα αυτά συμβαίνουν ήδη, διότι έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια σε ένα πρόγραμμα. Αυτά πρέπει να τα τιμήσουμε, ε, πρέπει να παρακολουθούμε ουσιαστικά το πρόγραμμα και κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχω τίποτα να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ, στηρίζω την έκθεση. Ευχαριστούμε τον Μίχαηλ ε, για δύο μόνο λεπτά, ενάμιση μάλλον. Κυρία Εγώ το Σεπτέμβριο με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Πακιστάν. Όντω ε, η έκθεση αυτή είναι πολύ καλή βάση συζήτηση. Θα καταθέσω τροπολογίες κυρίως σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται ακριβώς για μια χώρα που ε, ειλικρινά σκιαγραφεί αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Έχουμε και πάλι ε, στη χώρα αυτή μεγάλη επιρροή των πολύ φονταμενταλιστών Ισλαμιστών που έρχονται και από την ε, Σαουδική Αραβία. Ανέφερε το θέμα των σχολείων Μαντράσα ο εισηγητής. Εγώ ήρθα πεπισμένη ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πρέπει να κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση του βαθμού ε, σεβασμού και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ξέρουμε επίσης ότι στο Πακιστάν και σε όχι μόνο αλλά ε, και για μας ε, είναι καταστροφικό το θέμα της χρησιμοποίησης των μη επαδρομένων αεροσκαφών που χρησιμοποιεί ε, η ΙΠΑ στη χώρα αυτή. Υπάρχουν οι μειοψηφίες των γυναικών, των παιδιών που υποφέρουν, οι χριστιανοί. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει σχεδόν καθόλου με αυτούς και θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο φως. Εν πάση περιπτώσει θα καταθέσω τροπολογίες. Πολύ σύντομη κυρία Νίτς, πάρα πολύ σύντομα. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια κάποια ε, αναφορά στις φυσικές καταστροφές στο Πακιστάν, δηλαδή πλημμύρες, σεισμούς, διότι ξέρουμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα υποφέρουν από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Επίσης, το θέμα των εμπορικών συναλλαγών είναι σημαντικό. Και θα πρέπει να διαρωτηθούμε εάν τέτοιου είδους σχέσεις είναι μονόδρομος, αν εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι υποβάλλουμε αιτήματα, προσφέρουμε ε, ελάχιστα ζητώντας πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών λήγει στις 8 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Και περνούμε τώρα στο επόμενο θέμα. Uh, Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μέτα, εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου στην Αλβανία για την κατάσταση μετά τις εκλογές και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του Πρόεδρου μας κυρίου Μπρόκ που έπρεπε να συμμετάσχει στη διάσκεψη των Πρόεδρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην ανταλλαγή απόψεων και χαίρομαι πάρα πολύ που παρίσταται ο κύριος Μέτα εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας ε, αναπτύξετε τις δικές σας ε, παρατηρήσεις για την κατάσταση στην Αλβανία. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που με έχετε καλέσει στην ΑΦΕΤ σήμερα. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή την Αλβανία και την όλη διαδικασία προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη τη σταθερή που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι σήμερα η ΑΦΕΤ έχει υιοθέτησε το ψήφισμα για την Αλβανία αντικατοπτρίζει την προσοχή σας προς την περιοχή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ ρεαλιστική προσωρινή έκθεση και διότι έχει χορηγήσει το καθεστώς υποψήφια χώρα στην Αλβανία. Νομίζω ότι τώρα έχουμε περάσει σε ένα πάρα πολύ θετικό βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που αντικατοπτρίζεται από τις πολιτικές αλλαγές και τις εξελίξεις των τελευταίων μιλών μετά από πάρα πολλούς καυτούς μήνες και χαμένες ευκαιρίες κατορθώσαμε τελικά να βρούμε μια συμβαστική λύση για να μπορέσουμε να λύσουμε και όλα τα θέματα νοθομετικά τα οποία ήταν εκρεμή και να ανταποκριθούμε στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν οι εκλογές του Ιουνίου Δημοκρατικές, ελεύθερες και σημαίνουν ότι γίνεται τώρα με ευρωπαϊκό τρόπο το, η, ακολουθείται με ο, δημοκρατικό τρόπο η όλη δημοκρατική διαδικασία. Από τότε που στάθηκε το νέο μας δημοκρατικό κοινοβούλιο έχουμε ένα θετικό πολιτικό κλίμα, το καλύτερο τα τελευταία τρία χρόνια. Οι πάντες θα πρέπει να επενεθούν για αυτή την προσπάθεια και εδώ φαίνεται πόσο ε, πολύ έχει επηρεάσει την όλη κατάσταση η ευρεία συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν σε όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, στην Ολομέλεια και στις διάφορες κοινοβουλευτικές μας αντιπροσωπείες στο ε, εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση δεν έχει πολλές έδρες, πάντα είναι παρούσα σε όλες τις ε, αντιπροσωπείες στο εξωτερικό. Ως πρόεδρος της Βουλής, με μεγάλη ευχαρίστηση σας λέγω ότι από τότε που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας τον Σεπτέμβριο, κυρίως εστιάζουμε την προσοχή μας στην εξασφάλιση ε, της καλύτερης δυνατής πολιτικής συνεργασίας σε ανώτατο επίπεδο, πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και στους τελευταίους τρεις μήνες είδαμε να υπάρχει καλύτερη ποιότητα στις συζητήσεις μεταξύ πλειοψηφία και αντιπολίτευσης. Η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα μέτρα που λαμβάνονται είναι από τα κύρια θέματα που συζητώνται τους μήνες αυτού στο Βουλή μας. Πάρα πολλές ε, συναντήσεις, ακροάσεις ε, οργανώνονται και σήμερα λειτουργεί σωστά η Βουλή μας. Βοηθούμεθα από το νέο εσωτερικό μας κανονισμό πολύ που ψηφίστηκε με συνένεση τον προηγούμενο Μάιο έτσι όπως είχε απαιτήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι υπέρ του διαλόγου και όλοι πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε έναν επικοδομητικό πολιτικό διάλογο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις ε, ρυθμίσεις τις ε, πολιτικές, πράγμα που πρέπει να γίνει με ε, πνεύμα διαλόγου που να συμπεριλαμβάνει τους ε, πάντες ώστε να μπορέσουμε όλοι να συνεισφέρουμε στην δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του Κοινοβουλίου. Η επικοδομητική δουλειά η οποία γίνεται μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι ορατή και εφικτή. Τον επικεφαλής του συνταγματικού δικαστηρίου, τον εκλέξαμε πριν από 1,5 μήνα με συνεργασία και όλες οι πολιτικές δυνάμεις συνεισέφεραν. Τον προηγούμενο μήνα, για πρώτη φορά στο, στο δικό μας κοινοβούλιο, δημιουργήθηκε μια συμμαχία γυναικών ε, βουλευτών. Έτσι, η Βουλή μας ενέκρινε με ένα ψήφισμα για την ευρωπαϊκή ένταξή μας ζητώντα την κυβέρνηση και στα άλλα θεσμικά όργανα να επιταχύνουν το βήμα ώστε να ανταποκριθούν στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητήσαμε σε όλους να υπερψηφίσουν την προσχώρηση της Αλβανίας. Πιο πρόσφατα, έχοντας ακούσει όλες τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και όλων, ψηφίσαμε υπέρ της προσ των δικαιωμάτων των παιδιών στην Αλβανία, αποτέλεσμα εργασίας δύο επιτροπών και συνεργασίας πολιτικών ομάδων μετά από διαβούλευση της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων που εργάζονται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να σας πω ότι η ολομέλειά μας ποτέ δεν έχει διακοπεί εξαιτία πολιτικών διαφιλονικιών και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα και όλοι θα συνεργαζόμαστε με πνεύμα ε, συμπερίληψης και όχι αποκλεισμού. Θέλουμε να συνεχίσουμε δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε τρομερά σημαντικά βήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα τον δικαστικό και τον διοικητικό. Και η δική μας η δέσμευση και η δική μου προσωπικά θα είναι να συμπεριλαμβάνουμε τους πάντες στο ότι γίνεται στην χώρα μας. Αρχίσαμε με την εκπόνηση ενός σχέδιου δράσης ώστε να μπορούμε έγκαιρα και αποδοτικά να ασχοληθούμε με όλα τα εκκρεμή θέματα τα οποία έχουμε. Πράγμα που θα μας επιτρέψει να είμαστε αποδοτικοί και να εργαζόμαστε με διαφάνεια. Όπως ίσως επίσης ε, γνωρίζετε, έχουμε και μια νέα σχέση συνεργασίας με τον Ombudsman και έχουμε πει ότι όλες οι συστάσεις και οι εκθέσεις που συντάσσονται από αυτό το θεσμικό όργανο τόσο σημαντικό θα συζητηθούν και θα ληφθούν υπόψη κάθε φορά που ψηφίζουμε ένα σημαντικό νομοθετικό θέμα. Ο Ombudsman, όπως ξέρετε, επίσης επιτυχώς ε, έχει ασχοληθεί και με το θέμα των Ρωμά και έχει ε, κάνει όλη την κοινωνία να συνειδητοποιήσει τα προβλήματα που υπάρχουν. Οι συστάσεις τους έχουν τελικά υποβληθεί ώστε να μπορέσει να επιληθεί κυρίως το θέμα της στέγασής τους και η χορήγηση οικονομικής βοήθειας, πρόσβαση στην παιδεία για την ένταξή τους στην κοινωνία μας. Επίσης πιστεύω ότι η συνεργασία με ανεξάρτητα θεσμικά όργανα και με την κοινωνία των πολιτών θα μας βοηθήσει να ενισχυθούμε ακόμη περισσότερο σε επίπεδο της Βουλής. Εμείς θα πρέπει επιδείξουμε επίσης πνεύμα διαφάνειας όταν εκπονούμε νομοθετικές πράξεις που θα αποτελέσουν τη βάση καλύτερης ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των Η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ομάδων ε, συμφερόντων και η συνεργασία με διεθνείς εταίρους είναι κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να αποδείξουμε την αξιοπιστία των θεσμικών μας οργάνων. Η υποστήριξη λοιπόν προς όλα τα θεσμικά όργανα της χώρας μας είναι σημαντική. Χαίρομαι διότι στις 29 Οκτωβρίου η κοινοβουλευτική ε, Επιτροπή Σταθεροποίησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλβανίας συνεδρίασε και εξέδωσε διάφορες επικοδομητικές συστάσεις. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στα Τύρανα και μας βοηθήσατε να φτάσουμε σε συμβαστικές λύσεις όσον αφορά τέτοιου είδους συστάσεις. Άρχισε επικοδομητικός διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού μας και του Επιτρόπου, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε εφικτά αποτελέσματα και να εξασφαλίσουμε το ότι θα μπορέσουμε να ε, φέρουμε σε πέρα τις προτεραιότητες έτσι όπως τις έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δέσμευσή μας είναι να μπορέσουμε να επιταχύνουμε το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα κριτήρια ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε όσο το συντομότερο γίνεται τον ε, ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχουν περάσει μόνο τρει μήνε από τότε, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει μεγάλε προσπάθειε για να αποδείξουμε ότι είμαστε κράτο δικαίου. Καταπολεμούμε την διαφθορά. Ο σχετικό συντονιστή έχει διοριστεί και εκπονεί τη νέα στρατηγική κατά της διαφοράς. Νέα πακέτα μέτρων κατά της διαφορές συζητώνται και λαμβάνουμε πολύ αυστηρά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε κυρίως την ε, υψηλού επίπεδου αν θέλετε διαφορά με δίμευση των περιουσιακών στοιχείων ε, των ε, εμπλεκομένων σε περιπτώσεις διαφοράς. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επίσης ανέλαβε δράση και πειθαρχικά μέτρα κατά των δικαστών που παρακολύουν την ομαλή ε, διεξαγωγή των διαδικασιών καθώς και μέτρα κατά των παρανόμεν δράσεων που λαμβάνονται για να μην εφαρμοστεί σωστά ο νόμος από τις εθνικές διοκτικές αρχές. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και η Γενική Εισαγγελία συνεργάζονται για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν οποιαδήποτε μορφή εγκληματικότητας. Επίσης, οι διοκτικές αρχές ε, συνεργάζονται και με την, ε, σε όλα τα επίπεδα της αστυνομία για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας για να καταπολεμήσουμε τέτοιου διστάριστα φαινόμενα. Και τις επόμενες μέρες προβλέπεται μια συντονιστική συνευρίαση με τους ε, Ευρωπαίους εταίρους μας για την καταπολέμηση εγκληματικών πράξεων, εμπορία ανθρώπων και άλλου τέτοιου είδους παράνομες πράξεις τις οποίες θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Επίσης θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα των Αλβανών που ζουν σε άλλες χώρες και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν. Τι πιστεύουμε σε μια ευημερία της περιοχής και θέλουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας. Δεν θεωρούμε ότι η απόδοση του καθεστώτος ε, υποψηφίας προς προσφόρηση χώρας είναι το τελικό σημείο. Ε, θεωρούμε ότι είναι ένα ορόσημο το οποίο θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο ε, ευθυνών και υποχρεώσεων για την Αλβανία. Επίσης, επιτρέψατε μου να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο σημαντικό. Ενώ, ε, σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου το Δεκέμβριο, θα συνεχίσουμε ταχαίως τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ξεκινήσαμε. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται εις όφελος της Ευρώπης, αλλά για να υπηρετήσουν το, εξυπηρετήσουν το καλό των πολιτών μας. Και στο βαθμό που συνδέονται με την χορήγηση της ε, υποψηφιότητας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό σημαίνει μια περαιτέρω ενθάρρυνση για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μέτα για την έκθεσή σας και την πολύ θετικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα σας τους τελευταίους μήνες. Και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους. Πρώτος είναι ο κύριος Κούκαν, ο οποίος είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας ε, ε, για την Αλβανία. Ε, είναι πολύ καλό που σας βλέπουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Κάνατε μια πολύ καλή ομιλία και είναι δύσκολο να μέμψω κάτι στην ομιλία σας γιατί αποστήλατε όλα τα ορθά πολιτικά μηνύματα και θα ήθελα πραγματικά να σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας στην κατεύθυνση που εκφράσατε, που διατυπώσατε εσείς μάλλον στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Ο καθένας εδώ εκτιμά πραγματικά ε, τη νέα ε, θετική ατμόσφαιρα στη, στη χώρα σας ξεκινώντας από τις εκλογές, την αποδοχή της ΣΥΤΑΣ ε, εκ μέρους της προηγούμενης κυβέρνησης και την ε, ταχεία μετάβαση της κυβερνητικής ε, εξουσίας καθώς και τα βήματα που δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο στην παρούσα συγκυρία λειτουργεί καλά, κάτι ποτέ συμβαίνει, δεν είναι εξασφαλισμένο πάντοτε στην Αλβανία. Θα ήταν εσφαλμένο να πούμε ποιος συνέβαλε περισσότερο προς αυτή τη νέα θετική πλέον ε, κατάσταση. Αυτό το οποίο ζητάμε από εσά είναι το εξής. Ε, εμείς ε, χρειαζόμαστε περισσότερες αποδείξεις στο μέλλον ότι πραγματικά έχει δρεωθεί αυτή η νέα κατάσταση γιατί θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω. Συμφωνώ ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν θαύματα σε μερικούς μόνο μήνες και δεν νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά ρεαλιστικό να απαιτήσουμε από εσά να κάνετε θαύματα αλλά θα πρέπει να δείξετε ε, πράγματι να αποδείξετε ότι υπάρχει αυτή η νέα θετική στάση, υφίσταται και μπορεί να λειτουργήσει ως βάση οικοδόμησης ε, για άλλα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει αυτή, υφίσταται αυτή η τάση στην Αλβανία Έχουμε το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε στις 27 Νοεμβρίου. Πολύ καλό ψήφισμα, ακριβώ όπως και η ομιλία σας. Και πραγματικά η ημερήσια διάταξη της ολοκλήρωσης είναι πολύ σωστή και καταδεικνύεται όλα τα σημεία τα οποία είναι τα προπατούμενα της ε, ολοκλήρωσης. Ε, της ένταξης. Ε, και το ψήφισμα καταρτίστηκε με τη συμμετοχή της κυβέρνησης, των κυβερνητικών δυνάμεων, αλλά και της αντιπολίτευσης, η οποία ε, συνέβαλε θετικά. Άρα πρόκειται εδώ για μία άλλη απόδειξη ότι τα πράγματα αλλάζουν και κινούνται ταχαίως. Δόξα το Θεό. Όταν λέμε ότι θα πρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας και θα πρέπει να μας κομίσετε και άλλες νέες αποδείξεις. Το λέμε επειδή ε, ε, ε, εγώ πραγματικά σας πιστεύω και θέλω να σας δώσω μια ευκαιρία. Δεν είμαι αισιόδοξο, δεν είμαι απολύτως αισιόδοξο. Πιστεύω ότι εσείς προσωπικά μπορείτε να διαδραματίσετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ένταξη της Αλβανίας. Το κάνατε άλλωστε και στο παρελθόν και θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές συμμερίζονται την άποψή μας. Και υπάρχουν ε, κάποιοι, κάποιες άλλες χώρες που λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες από την Αλβανία που αιτούν άσυλο. Ε, τα πράγματα σχέση με τις ε, θεωρήσεις δεν είναι και τόσο καλά τελευταία και ίσως θα πρέπει να κάνετε κάποιες θετικές αλλαγές, διορθώσεις εδώ πριν από τις εκλογές, γιατί θα πρέπει να έχετε συνείδηση αυτή της κατάστασης και να μην δώσετε ευκαιρία στην πλευρά που δεν επιθυμεί την ένταξη της Αλβανίας να έχει στα χέρια της κάποια του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενθαρρυντική παρέμβαση. Ο επόμενος ομιλητής είναι μόνιμος συγητής για την Αλβανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω εδώ. Κυρίως ε, σήμερα που έχουμε και ευχάριστα γεγονότα. Το ψήφισμα για την Αλβανία είναι αρκετά θετικό ε, και νομίζω όπως ξέρετε ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα στην Επιτροπή μας. Μόνο μία αποχή είχαμε και όλοι οι άλλοι αποδέχτηκαν το ψήφισμα. Την επόμενη εβδομάδα το ψήφισμα θα κατατεθεί στην Ολομέλεια. Επιμείναμε επ' αυτού για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε σαφή θέση του Κοινοβουλίου επί του θέματος και θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια πριν ληφθεί η τελική απόφαση στο Συμβούλιο. Κανείς μας βέβαια δεν ξέρει τι θα συμβεί στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες εικασίες από πλευράς ε, διπλωματικών κύκλων, αλλά θέλω να ελπίζω ότι το μήνυμα του Κοινοβουλίου θα φτάσει στο Συμβούλιο και αυτό θα αποβεί προς όφελος της χώρας σας. Και αναφέρομαι όχι μόνο στο μήνυμα του Κοινοβουλίου. Είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται βλέπουν ότι υπάρχουν εξελίξει στην Αλβανία, ένας νέος τρόπος σκέψης και πόσο σημαντική έχει γίνει η λέξη συμβιβασμό. Όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά, μιλάγαμε για συνένεση. Εγώ είχα πει η λέξη συνένεση είναι κακή γιατί έχει κάποιες κακές αποχρώσεις, ε, κυρίως για μας που ε, ζήσαμε στις, ε, στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία. Συμβασμός είναι η καλύτερη λέξη, αυτή μας άρεσε. Και προφανώς, από ό,τι φαίνεται, επιτύχατε έχετε ε, την ε, αντιπολίτευση πλέον ε, στη χώρα σας. Υπάρχουν βέβαια και πολλά θέματα που πρέπει να επιληθούν, η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, η φτώχεια, η οργάνωση της διοίκησης και πολλά άλλα. Δεν έχω όμως καμία απολύτως αμφιβολία ότι οι Αλβανοί θα τα λύσουν αυτά τα προβλήματα και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Βεβαίως και δεν μπορούν να γίνουν θαύματα ε, μέσα σε λίγους μήνες ε, έτσι απλά. Ε, είδαμε ας πούμε τι έγινε στα Τύρανα που άνθρωποι κατέβηκαν κατά της πυρηνικής δύναμης και κυρίως στη Συρία. Ε, και η κυβέρνηση άκουσε την άποψη των ανθρώπων. Αυτό εγώ θα το χαρακτηρίζα θαύμα γιατί πραγματικά είναι ένας νέος τρόπος ε, σκέψης. Η χώρα λοιπόν έχει επιτύχει πάρα πολλά. Εμείς προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε στο βαθμό του δυνατού και είμαι Βεβαίως πιστεύω ότι τα πράγματα ακολουθούν το σωστό δρόμο και θα συνεχίσουν ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο καθένας ε, εκτελεί αυτό που του αναλογεί. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρούτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρα να σας καλωσορίσω και να συνεχίσω με αυτό το θετικό πνεύμα. Όπως μπορείτε να δείτε σήμερα και στο δικό μας ψήφισμα και στην ε, ψηφοφορία υπάρχει υποστήριξη αν συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση η Αλμπανία και θα συνεχίσει να υπάρχει υποστήριξη όχι μόνο από τους σοσιαλιστές αλλά και από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Αναφέρατε τη λέξη inclusiveness που είναι συμπερίληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, συμπερίληψη στο Βουλή σημαίνει συνεργασία κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το είδαμε και πριν από τις εκλογές και τώρα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να συμπεριλαμβάνονται όλοι στη πνεύμα συνεργασίας ό,τι γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει με την κοινωνία των πολιτών, με τον λαό σας, διότι η Βουλή οι εκπρόσωποι της Βουλής εκλέγονται από τον λαό. Άρα είναι πάρα πολύ καλό να διαβουλεύεστε όχι μόνο τις άλλες πολιτικές ομάδες, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Και βεβαίως εδώ δεν μπορούμε να πούμε ε, ότι πρόκειται για θαύμα, αλλά για πολλά θετικά σημεία, πολλά συν τα οποία προστίθεται στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριλαμβάνει σε ό,τι κάνει και την ε, κοινωνία των πολιτών. Πολύ καλά επιχειρήματα είναι αυτά. Χρειάζεται συνεργασία, αναφέρεται και το σχετικό ψήφισμα. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ, όπως είπατε, γνωρίζετε τι ακριβώς πρέπει να γίνει στο δικό σας το γήπεδο είναι το μπαλάκι, πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, διοικητικοί και άλλες, για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τη διαφθορά και το οργανωμένο ε, έγκλημα, πράγμα το οποίο δεν είναι σημαντικό μόνο για την προσχώρησή σας, αλλά για την ε, σωστή λειτουργία της αλβανικής κοινωνίας και για την ε, οικονομία σας. Θα πρέπει λοιπόν επικεντρώστε τις προσπάθειές σας και στο πώς θα λειτουργήσει σωστά η οικονομία σας. Βρίσκεστε σε καλό δρόμο, έχετε πολλές δυνατότητες. Και έχω εμπιστοσύνη ότι θα δημιουργήσετε, θα ε, μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε σωστά όλες αυτές τις δυνατότητες που έχετε για να προχωρήσετε. Επίσης θα ήθελα να ε, αναφέρω το εξής. Υπάρχουν ευκαιρίες. Η χώρα σας και εσείς στη Βουλή σας θα μπορέσετε να εστιαστείτε στην ε, ε, συνεργασία την περιφερειακή της δικής σας περιοχής. Έχετε το Μαυροβούνιο δίπλα που διαπραγματεύει, σύντομα θα αρχίσει η Σερβία, υπάρχει μεταξύ ε, Πρίστινα και Βελιγραδίου διάλογος, εκλογές στο Κωσυφοπαίδιο, πολλά πράγματα γίνονται στην περιοχή. έχετε λοιπόν την πολύ καλή ευκαιρία να συνεργαστείτε σε περιφερειακό επίπεδο και εσείς ως πρόεδρος της Βουλής μπορείτε να διαδραματίσετε θετικό ρόλο στον τομέα αυτό και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα σας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως Το καθεστώς της υποψήφιας χώρας στην Αλβανία είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι το σημείο τερματισμού σας. Είναι κατά κάποιο τρόπο η αρχή προς ένα νέο στάδιο και ότι οι δυσκολίες υπάρχουν εσωτερικά θα πρέπει να επιληθούν και με το πνεύμα της διαπραγμάτευσης όλο περισσότερο να προχωρείτε προς την εξέβριση λύσης. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν σας χορηγηθεί αυτό το καθεστώς, τόσο καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατσίν, τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, ε, κύριε πρέσβη, χαίρομαι που ξαναβρίσκεστε εδώ με μια νέα ιδιότητα, αλλά το να είναι κανείς πρώης βουλής είναι το δεύτερο σημαντικότερο αξίωμα σε ένα κράτος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η θέση σας. Επειδή σας γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, ξέρω ότι δεν θα είστε απλώς παρατηρητής, αλλά θα είσαστε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της αλβανικής κοινωνίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρξει εκδημοκρατισμός. Ε, η κατάσταση τώρα είναι μεταβατική. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Εθνικού Κοινοβουλίου, όπως και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να είναι πιο αποτελεσματική η ευρωπαϊκή θεσμή και πιο κοντά στους πολίτες. Νομίζω λοιπόν ότι ο δικός σας ρόλος, ο ρόλος του Προέδρου της Βουλής είναι ιδιαίτερα σημαντικός για να κατανοήσουν οι άνθρωποι πώς και τι πρέπει να γίνει η κατάργηση των ε, αποκλεισμών ξεκινάει από το Κοινοβούλιο. Η αντιπολίτευση οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της, όχι μόνο να αντιπολιτεύεται και να κάνει φασαρία. Η Αλβανία έχει χάσει πάρα πολύ καιρό. Ε, Εμεί δείξαμε υπομονή και τώρα έχετε επανέλθει. Σας παρακαλώ λοιπόν να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια και είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε όλα αυτά που αναφέρθηκαν σήμερα εδώ. Αυτά που είπατε στην αρχή ήταν πραγματικά εξισορροπημένα και πολύ ευχάριστα για τα αυτιά μας. Ε, αυτά περιμέναμε. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Από την άλλη, Θέλω να σας στηρίξω στις προσπάθειές σας με βάση τις προηγούμενες θέσεις που είχατε. Ξέρετε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, με τους γείτονες. Ε, ε, χρειαζόμαστε επιγόντως να γίνει κάτι με τη Μακεδονία, τον άμεσο γείτονά σας. Υπάρχει εκεί μια σημαντική αλβανόφωνη μειονότητα και αυτή λοιπόν πρέπει να είναι επικοδομητικοί παίκτες. Μιλάω για τον εκδημοκρατισμό της Μακεδονίας, όχι για την ένταξή της, γιατί αν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές εκδημοκρατισμού δεν θα μπορέσει η Μακεδονία να προχωρήσει δεν θα υπάρξει συνέχεια. Έτσι λοιπόν πρέπει να τους ε, επαναφέρουμε στην πραγματικότητα και πιστεύω ότι και εσείς ε, μπορείτε να τους ε, βοηθήσετε για να κάνουν και εκείνοι ό,τι μπορούν. Βλέπουμε λοιπόν την Αλβανία ως ένα ιδιαίτερα επικοδομητικό παίκτη. Προς το παρόν ήμασταν Γκόρι, Πογκορίτσα Πρίστινα, ένα πολύ καλό ε, τρίγωνο. Θέλουμε να προσθεθούν και τα τύρανα ε, σε αυτό το σχήμα για να υπάρξουν ε, θετικές αλλαγές στην περιοχή. Χαίρομαι λοιπόν που ήρθατε εδώ και ελπίζω να έρχεστε πιο συχνά γιατί αυτό ε, θα ήταν θετικό όχι μόνο για σας αλλά και για μας. Για μας ως ε, Επιτροπή και για τον θεσμό μας γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς λέει ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Πρόεδρε, τώρα δικό σας ο χρόνος μέχρι <laughs> να ολοκληρωθούν οι εργασίες μας που είναι δηλαδή πέντε λεπτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τον κύριο κοκάν, τον κύριο Βούλκανιτς, τον κύριο Λούτσεκ και τον κύριο Κατσίν για τα σχόλια τους, για τις παρατηρήσεις τους, για την ε, μεγάλη υποστήριξή σας προς ε, την Αλβανία και την όλη διαδικασία προσχώρησης της χώρας μας. Ενεργά επίσης υποστηρίξατε το ψήφισμα που υιοθέτησε η Επιτροπή σας είσαστε πιο επικριτικοί στο παρελθόν γιατί αντιμετωπίζαμε περισσότερα προβλήματα. Τώρα έχετε πιο θετικό πνεύμα προς εμάς, διότι η Αλβανία τους τελευταίους μήνες κατέληξε σε θετικά αποτελέσματα. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι ομόφωνα το τελευταίο ψήφισμα που υιοθετήσαμε στη Βουλή μας πρέπει να σας πω ότι προήλθε από την αντιπολίτευσή μας που ήταν πολύ ενεργός και με την συνεργασία μεταξύ όλων ημών μπορέσαμε σε πολλές περιπτώσεις να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για όλα τα πολιτικά κόμματα και τις δυνάμεις είναι κοινό στόχος η ευρωπαϊκή μας προσχώρηση και στις τελευταίες όλοι ψήφισαν με μεγάλο ε, πνεύμα ευθύνης καταρρύπτοντας τους εθνικισμούς και υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας. Ξέρετε ποια είναι τα προβλήματά μας και όπως γνωρίζετε συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ποια είναι η προβληματική. Προσπαθούμε και με διμερείς συνεργασίες ή με πολυμερή συνεργασία να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Και βεβαίως θέλουμε κάθε μέρα να είμαστε αποδοτικοί και να εργαζόμαστε στεναρά. Και όχι μόνο μέχρι την ημέρα που θα παρθούν οι αποφάσεις από το αλλά και πέραν. Διότι πρώτα απ' όλα έχουμε αίσθημα ευθύνης προς τους πολίτες μας και θα συνεχίσουμε προς την σωστή κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε τις πέντε συστάσεις. Έχουμε επικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αλβανίας. Συνεχίζουμε ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε να επιτευθεί πρόοδος και να μπορέσει όλη αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η δύναμη των ε, μεταρρυθμίσεων που πνέει σε όλη την περιοχή μας βοηθά να προχωρήσουμε. Βλέπουμε τι ακριβώ συμβαίνει και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, με το Κωσυφοπέδιο, με το Μαυροβούνιο. Θα συνεχίσουμε να είμαστε ακόμη και πιο δυναμική. Πριν από δύο μήνες συζήτησα με τον πρόεδρο της Βουλής Μαυροβουνίου. Εδώ και δύο μήνες δημιουργήθηκαν ε, στην ε, δική τους Βουλή ομάδες φιλίας με μας και εμείς θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίσης με την ε, Σερβία θέλουμε να αναπτύξουμε σχέσεις φιλίες. Το θέμα της εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας είναι σημαντικό διότι έτσι θα βελτιωθεί η εικόνα, αν θέλετε, όλη τη περιοχή προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω προς του επενδυτέ. Γιατί είναι πρωταρχική σημασία για μα να αλλάξουμε ε, πλήρω την εικόνα για την περιοχή μας. Ακόμη δεδομένου ότι υπάρχουν διάφορες ε, παλιές αντιλήψεις και κάποια άλλη τα προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε, υποφέρουμε από αυτό το γεγονός. Θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Τώρα, όλες οι χώρες και εμείς το ίδιο θέλουμε να σταματήσουμε την εμπορία ανθρωπίνων όντων και να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Και προσπαθούμε. Αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει μια θετική εικόνα για την περιοχή μας, όχι μόνο μας επειδή να προσεγγίσουμε και να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ενθαρρύνει και τους επενδυτές να έρθουν στην περιοχή μας όλο και περισσότερο στο εγγύς μέλλον. Και αυτό είναι πρωταρχική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, για την ανάπτυξη τον ε, του λαού μας και την βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση, σας διαβεβαιώνω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας και προς αυτή την ε, θετική κατεύθυνση την οποία έχει λάβει η χώρα μας μετά τις εκλογές της 21ης Ιουνίου. Αυτές είναι δεσμεύσεις και προαρταρχικές προτεραιότητες για μας, όχι μόνο λόγια, θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όπως σας υπογράμμισα και πριν, η ευρωπαϊκή μας ένταξη είναι ένας εθνικός στόχος για τη χώρα μας. Υπολογίζουμε στην ε, υποστήριξή σας πολύ για το μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε... Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο συνάδελφος, αυτές οι θετικές πολιτικές εξελίξεις θα πρέπει να διαρκέσουν και να υπάρξει πολιτική συνεργασία. Το πνεύμα πολιτικής συνεργασίας θα πρέπει να ισχύσει και μελλοντικά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις προσπάθειές σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε εδώ και το τελευταίο σημείο της πρωινής συνεδρίασης. Καλή σας ε, όρεξη.